Bonjour. Καλημέρα. Υπάρχει απαρτία για να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Έχουμε μια σημαντική ψηφοφορία. Πρόταση προγράμματος υποστήριξης στις μεταρρυθμίσεις. 22 Νοεμβρίου 2018 Επιτροπή μας ενέκρινε τη θέση της με 21 ψήφους υπέρ και 4 ψήφους κατά. Όμως ε, η μεικτή Επιτροπή ΕΚΟΝ και, και Προπολογισμού δεν ψήφισε ποτέ την έκθεσή της. Ε, δεν ολοκληρώθηκε λοιπόν ποτέ αυτός ο φάκελος και γι' αυτό αναλάβαμε εκ νέου αυτόν τον φάκελο τώρα εδώ στην ε, σε αυτή τη θητεία. Οι συντονιστέ συζήτησαν το ζήτημα αυτό την προηγούμενη, προηγούμενο μήνα και είπαμε ότι θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε το φάκελο χωρίς τροποποίηση. Έτσι λοιπόν σήμερα έχουμε μια διαδικαστική ψηφοφορία χωρίς να υποβάλλεται κάποια νέα γνωμοτότηση και χωρίς ε, ψηφοφορία επιτροπολογιών. Ο νέος εισηγητής είναι ο αντιπρόεδρος μας, ο Κριστάν Γκινέα. Θα του δώσω το λόγο, εφόσον το επιθυμεί, ιδάλλως θα περάσουμε ε, απευθείας στην ψηφοφορία που θα είναι μία και μόνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. μια και είναι η ίδια ακριβώς νομοδότηση με αυτή της προηγούμενης επιτροπής, δεν υπάρχει λόγος να πω κάτι περισσότερο. Μάλιστα, πολύ ωραία, ευχαριστώ. Έχετε όλοι τις κάρτες σας. Μπορούμε λοιπόν να ψηφίσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται λοιπόν η έκθεση με 19 ψήφους υπέρ, 6 κατά και καμία αποχή. Συνεχίζουμε τις εργασίες μας. Ανταλλαγή απόψεων με την EuroCity, που είναι η βασική οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών που εκπροσωπεί τις πόλεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο δημιουργήθηκε το 1986 και συμμετέχουν σε αυτήν την ε, οργάνωση 140 από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης και βεβαίως εδώ έχουμε την προοπτική, την αμυγός αστική ε, για τη θέσπιση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Οι εργασίες της οργάνωσης θα μας παρουσιαστούν από ένα από τα μέλη της Εκλεστικής Επιτροπής της, το Ματίας Ντεκλέρκ, τον οποίο καλωσορίζω πρόκειται για τον Δήμαρχο της Γάνδης και βεβαίω να θυμίσω ότι ο Φρανσό Μιτεράν είχε επισκεφθεί τη Γάνδη, όλοι τη θυμούνται διότι είχε κάνει και μια ιδιαίτερη δήλωση τότε, είχε πει ότι η Γάνδη είναι η πιο γνωστή άγνωστη πόλη κατά κάποιο τρόπο. Μετά την παρουσίαση του κ. Ντεκλέρκ θα δώσω το λόγο στους βουλευτές για τα σχόλιά τους, τα ερωτήματά τους θέλησα να καλωσορίσουμε την EuroCity εδώ ε, όσο γίνεται πιο σύντομα γιατί παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη μάχη που δίνουμε για να υπερασπιστούμε την περιφερειακή πολιτική και βεβαίως ε, για να συνεχιστούν οι εργασίες ε, της προηγούμενης θητείας σε σχέση με το, την αστική ατζέντα το Σύμφωνο του Άμστερνταμ. Ελπίζουμε λοιπόν σε αυτή τη θητεία να συγκεκριμενοποιηθούν μια σειρά από στρατηγικοί προσανατολισμοί. Το έχουμε πει πολλάκις σε αυτή την Επιτροπή. Είναι πολύ σημαντικό το αστικό διακύβευμα. 70% του ψηφιτού πληθυσμού της Ένωσης ζει στις πόλεις και εκεί επικεντρώνονται και οι προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει η Ένωση, ιδιαίτερα οι περιβαλλοντικέ. Για το θέμα λοιπόν του κλίματος, ε, στις πόλεις ε, παίζεται το παιχνίδι και για τα ζητήματα ενεργειακής μετάβασης και για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την περιφερειακή πολιτική, η αστική φτώχεια, και το θέμα βεβαίως της ένταξης των μεταναστών, των προσφύγων, ζητήματα τα οποία είναι στην ημέρα διάταξή μας. Κύριε Ντεκλέρκ, σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ρέτζη, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία ως ε, δήμαρχος της ε, Γάντης, πανέμορφης πόλης που είναι μόλις 50 χιλιόμετρα από εδώ. Προς τα αριστερά στο χάρτη. Και ως βασικό μέλος της EuroCities, ευχαριστώ λοιπόν για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσω το δίκτυο EuroCities. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που είμαστε ο πρώτος οργανισμό ε, που έχει προσκληθεί εδώ στην Επιτροπή στην αρχή τη θητεία σα για να σας παρουσιάσουμε τις απόψει μα για την αστική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μοιραστούμε μαζί σας τα οράματά μα, τις ανησυχίες μας και τις προτάσεις μας για το μέλλον της Ευρώπης. Διότι είμαστε πεπισμένοι ότι η Ευρώπη είναι κάτι καταπληκτικό, την αγαπάμε, αλλά και η Ευρώπη πρέπει να αγαπάει τι πόλεις τη διότι εκεί ζουν οι πολίτε τη ε, Ευρώπη χωρίς ε, πολίτες είναι Ευρώπη χωρίς πόλεις. Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω το EuroCities. Πρώτα απ' όλα είναι το ηγετικό δίκτυο πάνω από 150 ευρωπαϊκών πόλεων που συνεργάζονται για τη βελτίωση της ε, ζωής στα αστικά κέντρα. Θέλουμε οι πόλει στην Ευρώπη να είναι πραγματικοί εταίροι με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να δημιουργούν, ε, κύριε Πρόεδρε, αυτό, με αυτό το σκοπό ένα καλύτερο μέλλον και τι θέτουμε στο επίκεντρο της ανάπτυξη ε, για ε, πόλεις που να χαρακτηρίζονται από ευημερία, από άριστο οποιοδήποτε αποκλεισμού. Ξεκινάμε ε, σε μικρό μέγεθο. ξεκινήσαμε με έξι πόλεις πριν από 30 χρόνια, το 1996. Και τώρα έχουμε ξεπεράσει τις 140 σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα μέλη μας είναι πόλεις με πάνω από 250.000 πολίτες και περίπου 50 κομοπόλεις επίσης ανήκουν στο δίκτυό μας και όλοι μαζί ε, δυστυχούμε σε 130 εκατομμύρια πολίτες ε, σε 39 χώρες. Ως ε, δίκτυο πόλεων αγαπητοί συνάδελφοι έχουμε θέσει έξι στόχους για την επόμενη δεκαετία. Πρώτον, οι πολίτες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν, να λαμβάνουν Μέρο ε, σε κοινωνίες χωρίς αποκλεισμού, ε, σε ευημερίε κοινωνίες, ε, να ζουν σε ένα υγιέ περιβάλλον, να έχουν ζωντανού δημόσιους χώρους, να αντιμετωπίζουν παγκόσμιες προκλήσεις και εκ των τα τοπικά συμβούλια των πόλεων θα πρέπει να εργάζονται για το μέλλον και θα συνεργαστούμε όλοι αυτοί, όλοι μαζί για αυτούς τους μελλοντικούς στόχους, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις με ολιστικό τρόπο και ολοκληρωμένο. Πιστεύω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σταυροδρόμι όπου η δημοτικά συμβούλια θα πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται με ένα νέο τρόπο, καινοτόμο. Ε, δεν μπορείς να κάνεις τα πράγματα μόνο σου. Γι' αυτό το λόγο οι Ευρωπαίοι πολιτικοί όλοι εμείς απευθυνόμαστε προς εσάς και σας απευθύνουμε έκκληση να συνεργαστείτε μαζί μας. Αγκαλιάστε μας. Δείτε μας ως συνεργάτες για να επιτύχουμε ανώτερους στόχους. Για παράδειγμα, χαιρόμαστε που θα εφαρμόσουμε εμείς το Green Deal και που θα καταστήσουμε την Ευρώπη την πρώτη ε, ουδέτερη χώρα, ουδέτερη υπηρό όσον αφορά τον άνθρακα μέχρι το 2050. Έτσι συνεργαζόμαστε με φιλόδοξες πόλεις ε, σε αυτό το πλαίσιο. Όλοι μαζί λοιπόν θα μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε αυτή τη μεταβολή. Σήμερα οι πολιτικοί ηγέτες συναντώνται στη Μαδρίτη, στην COP25 για να συζητήσουν για το θάρρος που χρειάζεται και την τόλμη στις πόλεις. Δεν μιλάμε απλά, κάνουμε και πράγματα, δράμε πραγματικά. Αυτό είναι σημαντικό. Και με περηφάνεια έχω να πω ότι η δική μου πόλη, η Γάνδη, πρόκειται να λάβει το βραβείο των ΗΕ στη Μαδρίτη για την τοπική μας στρατηγική για τα τρόφιμα. Πολύ συγκεκριμένες τοπικές δράσεις που έχουμε υλοποιήσει για να μειώσουμε το ανθρωπικό μας αποτύπωμα. Πάμε πίσω στο δίκτυο γύρωσή μέσω διαφόρων φόρα και ομάδων εργασία και έργων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων. Προσφέρουμε σε πολλά, στα πολυάριθμα μας μέλη μια πλατφόρμα ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών. Οι κοινότητες εμπειρογνωμόνων μας και πολιτικών εκπροσώπων είναι μεγάλες ε, με ισχυρούς δεσμούς και συνεργάζονται ε, πέραν οποιονδήποτε τοπικών ε, διαφορών. Η συνεργασία μεταξύ των πόλεων παρέχει μεγάλες λύσεις στην Ευρώπη, οικοδομεί ικανότητες στις πόλεις και φέρνει αποτελέσματα απτά για τους πολίτες. Το EuroCities επίσης είναι η ενωμένη φωνή των ευρωπαϊκών πόλεων ε, μπροστά στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Θέλουμε οι σχετικές πολιτικές και οι σχετικοί κανονισμοί που σχεδιάζονται στο δικό σας επίπεδο, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αντιστοιχούν στην πραγματικότητα που ζούμε εμείς στις πόλεις μας. Έτσι οι κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν κάποιο νόημα για τους πολίτες μας και θα βελτιώνουν τις ζωές τους. Ως δημοτικές αρχές ε, εμείς αποτελούμε μια αποτελεσματική γέφυρα για εσάς μεταξύ των πολιτών και τη θεματολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε το επίπεδο διακυβέρνησης που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη. Η δουλειά μας ε, κινείται προς δύο κατευθύνσεις. Συνεργαζόμαστε με τα θεσμικά οργάνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως στρατηγική εταίρη για να αντιμετωπίζουμε κοινά ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των ε, ε, πολιτών μας και δεύτερον, υποστηρίζουμε τα Δημοτικά Συμβούλια για να ενισχύσουμε το σημαντικό ρόλο που παίζουν στην ευρωπαϊκή πολυεπίπεδη κυβερνητική δομή. Πιστεύουμε ότι αυτή η νέα εντολή αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία για μας και ευχαριστώ για την πρόσκληση για να γεφυρώσουμε, κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάμε να αναφέρουμε, να γεφυρώσουμε ε, το κενό μεταξύ Ευρώπης και Ευρωπαίων. Εγώ πιστεύω στην Ευρώπη, ο, πατέ, ο παππούς μου ήταν επίτροπος και γεννήθηκε το 27 και στην πόλη μας ε, μπήκαν οι Ναζί και πέταξαν τους κατοίκους της Γάνδης από τα σπίτια τους. Ε, το είδε αυτό ως παιδί, ήταν 17 ετών στις 6 Σεπτεμβρίου του 1944 όταν η Γάνδη ε, απελευθερώθηκε από τους Πολωνούς και τους Καναδούς και γι' αυτό το λόγο ανέκαθεν έλεγε ότι πρέπει να ε, λειτουργούμε ως Ευρώπη. Πρέπει να συνεργαζόμαστε όλοι μαζί για να μην ξαναγίνει πόλεμος. Και αυτή είναι η μεγάλη ιδέα ε, ε, στην οποία πιστεύουμε εμείς, η Ευρώπη. Η Ευρώπη όμως τώρα πρέπει να βρίσκεται πιο κοντά και στους πολίτες και στις πόλεις. Ήθελα να πω αυτή τη σημαντική ιστορία, κύριε Πρόεδρε. Οι Ευρωπαίοι λοιπόν ε, ηγέτες ε, και οι εθνικοί ηγέτες ε, και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο όλοι πρέπει να συνεργαζόμαστε για να επιτύχουμε την Πράσινη Συμφωνία, το Πράσινο Σύμφωνο, να ενισχύσουμε ψηφιακό, την ψηφιακή μεταβολή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τέλος να αναγνωρίσουμε τη ζωτική κρίσιμη σημασία συμβολή των πόλεων στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Και ε, αυτό είναι ένα από τα μηνύματα που προσπαθεί να προωθήσει το δίκτυο μας στο Eurocities με την νέα εκστρατεία. Τη βρίσκεται στο ίντερνετ 100 ημέρες, 100 τρόποι. 100 days, 100 ways. Μπορείτε να το βρείτε στο Google. Και τις πρώτες 100 ημέρες εργασίας της Νέας Επιτροπής στέλνουμε μηνύματα συγκεκριμένα από το δίκτυό μας προς τους Ευρωπαίους πολιτικούς, προς εσάς για να συνεργαστείτε μαζί μας ε, στις 12 ε, σημαντικότερες προκλήσεις. Τώρα πάμε στο αστικό θεματολόγιο, αγαπητοί συνάδελφοι. Το 2016, κατά την άποψή μας, ήταν σημείο καμπής για μας, για τις πόλεις, διότι το αστικό θεματολόγιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθιερώθηκε τότε ε, από την Ολλανδική Προεδρία. Ξεκίνησε το Μάιο του 2016 με το Σύμφωνο του Άμστερνταμ περιλαμβάνει μια δέσμευση των κρατών μελών, της Κομισιόν και των ε, Δήμων να δοκιμάσουν νέους τρόπους συνεργασίας για ε, να αντιμετωπίσουν κοινά προβλήματα. Η φιλοδοξία ήταν η βελτίωση των κανονισμών, της χρηματοδότησης και καλύτερη ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των πόλεων. Βασιζόταν μια κοινή συνεννόηση, μια κοινή κατανόηση της ε, σπουδαιότητας των αστικών κέντρων στην Ευρώπη. Και σήμερα το είπε και ο πρόεδρος, το 70% του ευρωπαϊκού πληθυσμού ζει σε αστικά κέντρα. 85% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης παράγεται σε πόλεις. 70% της ε, νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εφαρμόζεται σε πόλεις και το 70% των θέσεων εργασίας δημιουργούνται σε πόλεις. Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους πιστεύω. Τα τελευταία τρία χρόνια οι πόλεις υπήρξαν όχι μόνο κομμάτι της εργασίας τους, 12 θεματικούς τομείς, ε, κλιματική αλλαγή, ποιότητα του αέρα, ε, αστική ένδυα, ψηφιοποίηση, έπαιξαν και κυρίαρχο ρόλο σε αυτές τις εργασίες. Και πρόσφατα έχουμε δύο νέες ε, εταιρικέ σχέσεις για τον πολιτισμό και την ασφάλεια, οι οποίες μόλις ξεκίνησαν. Θα πρέπει να είμαστε σαφείς λοιπόν κυρίες και κύριοι. Η οικονομική στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπήρξε ζωτική σημασία για την υλοποίηση του αστικού θεματολογίου γενικότερα. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε να τα αναφέρουμε. Ποια υπήρξε η προστιθέμενη αξία μέχρι στιγμής, ποια είναι τα μαθήματα, τα διδάγματα που αποκομίζουμε. Η Ρουμανική Προεδρία εκπονήσε μια αξιολόγηση εμείς κάνουμε μια έρευνα στο δίκτυό μας και η Κομισιόν σύντομα πρόκειται επίσης να ε, δημοσιεύσει μια αξιολόγηση και μπορείτε να δείτε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες δηλώσεις ε, στις διαφάνειες. Γενικά, ε, η αξιολόγηση εκφράζει εκτίμηση για τις προσπάθειες που έχουν γίνει στο πλαίσιο του αστικού θεματολογίου υπήρξαν από τα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, σαφεί ε, συστάσει για τη βελτίωση τη ευρωπαϊκή πολιτική και τη χρηματοδότηση για τι πόλει. αλλά και εργαλειοθήκες και κατευθύντηρες γραμμέ για την αντιμετώπιση των αστικών προβλημάτων. Εντοπισμό ε, προβλημα... Ε, δεδομένων και κενών στις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να βελτιώσουμε τις πολιτικές της πόλης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και η αστική ατζέντα συνέβαλε σε πολλά θετικά αποτελέσματα στο κοινωνικό κλάδο. Για παράδειγμα, επηρέασε τις διαπραγματεύσεις για το ΆΜΕΦ, για τα Ταμεία Ασύλου, Μετανάστευσης και ε, προσφύγων ε, για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι η αστική ατζέντα ενίσχυσε το διάλογο μεταξύ πόλεων, κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε πολλούς τομείς πολιτικής. Έτσι αποτελεί τη βάση για μια ισχυρότερη, πιο πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χάρη στην ε, καινοτόμο και πειραματική της ε, φύση, ε, αλλά φυσικά υπάρχει και περιθώριο βελτιώσεων. Θα σας παρουσιάσω εδώ κάποιες ιδέες. Για να έχει νόημα το αστικό θεματολόγιο, τα αποτελέσματά του θα πρέπει να μεταφράζονται σε πολιτικές ευρωπαϊκές. Οι προσπάθειες θα χαθούν αν τελικά όλε αυτέ οι πληροφορίες δεν ενσωματωθούν ε, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο. Επίση, το αστικό θεματολόγιο χρειάζεται και ισχυρότερη δέσμευση, ειδικότερα από, κράτη -μέλη, από τα κράτη-μέλη και από τι Γενικέ Διευθύνσει τη Επιτροπή. Ο σκοπό για τον οποίο υπάρχει το αστικό θεματολόγιο είναι οι εθνικέ κυβερνήσει και οι κομισιόν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με τι πόλει, με του Δήμου, να συζητήσουν στο επίπεδο μια πολυεπίπεδη κυβερνητική προσέγγιση για το πώ θα επιλύσουν κοινά προβλήματα. Για να επιτύχουμε του στόχου του Πράσινου Συμφώνου είναι αναγκαία η παρουσία των πόλεων και των Δήμων. Μόνο με τη συμμετοχή των πόλεων και των δήμων μπορούμε να επιτύχουμε του σημαντικού στόχου του Πράσινου Συμφώνου. Και τέλος, η δέσμευση αυτή θα πρέπει να προέρχεται, να συνοδεύεται από χρηματοδοτικά μέσα τα οποία θα χρησιμοποιούνται πιο αποτελεσματικά. Προς το παρόν, ε, η βασικότερη υποστήριξη παρέχεται από εξωτερικού εμπειρογνώμονε, αλλά πιστεύουμε ότι θα μπορούσαν να επιτευχθούν πολλά περισσότερα αν οι εταίροι σε αυτή την αστική ατζέντα είχαν στη διάθεσή του ένα ευρύτερο φάσμα εργαλείων. σε αυτή τη θητεία λοιπόν της Κομισιόν του Κοινοβουλίου εμείς διακρίνουμε νέε δυνατότητες που μπορούν να ενισχύσουν την αστική διάσταση καθώς και τη δημοκρατική, το δημοκρατικό χαρακτήρα των πολιτικών. Η πολιτική συνοχή και τα σχετικά μέτρα μετά το 2020 θα παίξουν εδώ σημαντικό ρόλο. Έχουμε συνεργαστεί πολύ στενά για, στο επίπεδο αυτό με την Επιτροπή σας και πολλές από τις προτάσεις σας έχουν ληφθεί υπόψη. Ε, πολλές από τις προτάσεις μας έχουν ληφθεί υπόψη σε ε, προτάσεις που κάνετε εσείς και σας ευχαριστούμε. Αλλά ε, ό,τι προτείνει το Συμβούλιο για την πολιτική συνοχή, όπως και στις διαπραγματεύσεις του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, ε, οι εξελίξει εκεί μα φαίνονται λιγότερο θετικέ και ήθελα να το αναφέρω αυτό ω εκπρόσωπο του EuroCities, διότι ανησυχούμε ιδιαίτερα για τι πιθανέ περικοπέ ε, στον προπολογισμό. Τόσο δραστικές περικοπές θα είχαν ως αποτέλεσμα ε, αρνητικά, αρνητικές συνέπειες για τις δυνατότητες που παρέχονται πόλης. πόλεις. και εκεί θα αμφισβητηθεί η δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκπληρώσει τους στόχους που έχουν θεσπιστεί στις συνθήκες για ε, κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή. Ε, θα οδηγήσει σε λιγότερες επενδύσεις σε βασικούς στόχους. Πρέπει λοιπόν να μην ξεχνάμε το πόσο σημαντική είναι η εταιρική σχέση να ενισχυθεί, ούτως ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών δαπανών, κάτι απαραίτητο για την ανάπτυξη κρίσιμων και κατάλληλων λύσεων στις πόλεις. Απορρίπτουμε λοιπόν οποιαδήποτε προσπάθεια αποδυνάμωσης αυτής της αρχής. Αυτό ήθελα να πω επίσης, ε, κύριε Πρόεδρε, σήμερα. Ο νέος συντονισμός ε, του χάρτη της λειψίας ε, που Πιστεύουμε ότι θα ενισχύσει κάποιε αρχέ, όπως την ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη, για να αντιμετωπίσουμε περίπλοκα αστικά ζητήματα. Επίσης, ε, θα επισημανθεί ανάγκη χειραφέτησης των πόλεων για να αντιμετωπίσουν με παγκόσμιο τρόπο τοπικές προκλήσεις. Θα ήθελα να τονίσω το εξή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητά τρόπου, επαφή με του πολίτε και οι λόγοι φυσικά είναι πολύ καλή Είναι καλή αυτή η επιλογή. Οπότε σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνηση θα πρέπει να δράσουμε ούτω ώστε να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη στου πολιτικού μα θεσμού για να ενδυναμώσουμε το κοινά μας ε, δημοκρατικά έργα. Η συνεργασία με τις αστικές αρχές, με τις δημοτικές αρχές, σημαίνει συνεργασία με τους πολίτες. και οι πολίτε μα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο τη πολιτική σκέψη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το δικό μας δίκτυο, το EuroCities, μπορεί να υποστηρίξει την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επιτευχή όλων αυτών. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε στη, μαζί σα στη διάσκεψη για το μέλλον τη Ευρώπη, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα, που θα ξεκινήσει σύντομα με πρωτοβουλία τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αγαπάμε λοιπόν όλοι μα την Ευρώπη και εγώ αγαπώ την Ευρώπη, αλλά η Ευρώπη δεν έχει μέλλον χωρί του πολίτε και χωρί τι πόλει τη. Οπότε συνεργαστείτε με τι πόλει, με του πολίτε και με το γύρωσή τη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε Ντεκλέρκ, σας ευχαριστούμε για την τοποθέτησή σας την τόσο θερμή. Επιχειρηματολογήσατε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, αλλά και ευρύ τρόπο και θα ξεκινήσουμε αμέσως αυτήν τη συζήτηση. Ήθελα να τονίσω την ποιότητα των σχέσεων και την καλή συνεργασία που έχουμε με τη γραμματεία των Γυροσίτης και την ε, Γενική Γραμματέα κυρία Αναλίζα Μπόνη που την καλωσορίζω επίσης η Επιτροπή μας πάντοτε συνεργαζόταν πολύ καλά με την Eurocities και είμαι σίγουρος ότι θα ενδυναμώσουμε ακόμα περισσότερο τις σχέσεις μας. Έχετε δίκιο ότι η απάντηση στις παγκόσμιες προκλήσεις δεν μπορεί παρά να εξαρτάται, να περνάει από το τοπικό επίπεδο και εκεί είναι που πρέπει να προχωρήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Εδώ έχουμε τους εισηγητές και συνεισηγητές στα διάφορα θέματα διαπραγμάτευσης. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι απολύτως πεπισμένο για τη χρησιμότητα των εταιρικών αυτών σχέσεων και συνεργασιών και πρέπει να συνεχίσουμε προς την κατεύθυνση αυτή όσο θα χρειαστεί. Λοιπόν, θα ανοίξουμε τώρα τη συζήτηση και θα ακούσουμε την κυρία Ιζαμπέλ Καχμπελέης από τους ε, σοσιαλιστές. Θα μιλήσω πρωτογαλλικά, Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω. Σας περιμένω. Θα ευχαριστούσα πρώτα απ' όλα τον κύριο Ματίας Ντεκλέρκ για την εξαιρετική του εισήγηση και να καλασορίσω επίσης ε, την γύρωσή της. Εγώ προέρχομαι από το βορρά της Πορτογαλίας ε, Ξέρω πόσο το δίκτυο αυτό έχει δουλέψει καταπληκτικά και ξέρω ότι έχει επιφέρει απτές βελτιώσεις για τους κατοίκους, για τους πολίτες μας. Εγώ ήθελα να πω ότι ο νέος κύκλος πολιτικής που δεν μας αφήνει σε ισχύα ε, προβλέπει συμφωνίες ή τουλάχιστον είναι, βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση για την πολιτική συνοχής δεν πρόκειται μόνο για μια συζήτηση επί επενδύσεων. Μιλούμε για τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Ε, όπως πολύ σωστά είπατε, πολλοί από τους πολίτες αυτούς ε, ζουν στα αστικά κέντρα στις πόλεις που συνθέτουν την Ευρώπη και όπως επίσης σωστά είπατε, οι πόλεις αυτές, τα αστικά κέντρα ε, είναι ένα σύνολο από τεράστιες προκλήσεις για την χρηστή διαχείριση ε, των υδάτινων πόρων, για την συμμετοχή, την κοινωνική ένταξη των μεταναστών. Ε, χρειαζόμαστε μια ισχυρή πολιτική συνοχή, χρειαζόμαστε να υποστηρίξουμε την συνοχή, διότι τα πιο σοβαρά προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι ε, κρίσιμη σημασία για πολλές από τις πόλεις μας. Ήθελα να διαβιβάσω λοιπόν αυτήν την ανησυχία αλλά και τη δέσμευση αυτή από πλευρά μου. Γιατί όταν κινήσουν αυτέ οι διαπραγματεύσεις ε, ε, εμείς δεν θα μείνουμε ε, με τα χέρια δεμένα, θα συμμετάσχουμε ενεργά για να προστατεύσουμε το μέλλον των πολιτών μας. Έχω μία ερώτηση να σας κάνω. Η σχέση της πόλης με την Ήπεθρο, ο συσχετισμός των δύο αυτών πλαισίων ζωής και δραστηριότητας. Πώς το βλέπετε αυτό να κινείται για το μέλλον. Γιατί ο καθένας από αυτούς τους κόσμους έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα είναι δύο τελείω χωριστοί κόσμοι. Ε, ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Ο κύριος Νόβακοφ ε, για το ΕΛΚ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να συγχαρώ τον Δήμαρχο εγώ εντυπωσιάζομαι από τέτοιες πρωτοβουλίες όπως η γύρωσή της και ως ε, συνομήλικο σας περίπου χαίρομαι που βλέπω νεότερους ε, που συνεισφέρουν με ένα νέο όραμα, ένα νέο πνεύμα στην πολιτική ζωή και όταν αυτό εκδηλώνεται σε περιφερειακό επίπεδο είναι ακόμα πιο ελπιδοφόρο. Βρίσκεστε σε μια επιτροπή όπου αναγνωρίζετε όσο ο καλύτερος φίλος μάλλον των περιφερειών. Δίνουμε μάχη για την καλύτερη χρηματοδότηση των περιφερειών, την προστασία της πολιτικής συνοχής, των χρηματοδοτικών μέσων που μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας ε, στο μέτωπο της συνοχής. Και συζητούμε σε μια στιγμή όπου συζητούμε για το μέλλον της πολιτικής συνοχής μετά το 2020. Ήθελα λοιπόν να μας πείτε την άποψή σας. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτή η πολιτική συνοχής μετά από ένα χρόνο. Θα πρέπει να μείνει για τις πιο ιστερούσες περιοχές ή θα πρέπει να περάσει το επόμενο σκαλοπάτι να είναι εποφελής για όλες τις περιφέρειες και για τις πιο προηγμένες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος Αντρέη Λουκτή του Ρινιού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε, για την παρουσίαση. Πολύ χαίρομαι που βλέπω ότι υπάρχει ένας φορέας που εξασφαλίζει καλύτερη συνεργασία, πιο ευφυείς στρατηγικές, ε, πιο περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνε πολιτικές για τις πόλεις. Κάποιες τυχές που συνδέονται με κάποια από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα στην Ευρώπη. οι οποίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την διαθεσιμότητα κατοικιών στεγαστικού χώρου, είτε ιδιόκτητου είτε ενοικίαση. Και βλέπουμε ότι νέα νοικοκυριά, νέε οικογένειες δεν καταφέρνουν να ζουν στις πόλεις, αλλά στην περιφέρεια τους και σε αρκετά μεγάλη απόσταση. Που σημαίνει ότι χρειάζονται μεταφορές πολύ συχνά πρέπει να χρησιμοποιούν αυτοκίνητα, υπάρχει συνοστισμός με τη στάθμευση των οχημάτων αυτών, υπάρχει περιβαλλοντικός αντίκτυπος. Ε, ήθελα λοιπόν να μου πείτε αν έχετε συζητήσει το θέμα αυτό στην γύρωσή τη. σχετικά δηλαδή με την δημιουργία, την οικοδόμηση καλύτερων συνθήκων ε, στη μεταφορά από και προς την πόλη των ανθρώπων που κινούνται έτσι για να εργαστούν. Δηλαδή με τα μέσα μαζικών μεταφορών και ώστε να αποφεύγονται οι μετακινήσεις με το αυτοκίνητο. Σας ευχαριστούμε Αντρέ. Για το ID η Φραντσίσκα Ντονάτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα Ιταλικά λέει η ομιλήτρια στα Ιταλικά. Και εγώ θα συγχαρώ τον ε, κύριο Δήμαρχο της Γάνιδης για την σαφήνεια της τοποθέτησής του. Είμαι πεπισμένη ότι το δίκτυο EuroCities είναι πολύ σημαντικό και πολύ αποτελεσματικό στη δουλειά του. Λυπούμε που δεν είναι όλες οι μεγάλες πόλεις της Ιταλίας που συμμετέχουν στο δίκτυο αυτό. Πραγματικά θα προσπαθούσα να δεσμευθώ ώστε να συμμετάσχουν πολύ περισσότερες ε, τουλάχιστον από τις περιφέρειες ε, στις οποίες εγώ εξελέγην στη Σικελία. Σας συγχαίρω για τη δουλειά σας και σας εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ιζαμπέλ Μπεντζουμέα, αντιπρόεδρος της Επιτροπής αυτής, έχει το λόγο. Θα μιλήσω ισπανικά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Δήμαρχο της Γάνδης, που για μας ε, τους Ισπανούς είναι πολύ σημαντική. Ε, πολύ γιατί ο Κάρολος ο Πέμπτος εκεί γεννήθηκε, μεταξύ άλλων. Ε, ήθελα να εστιαστώ σε ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό και σχετίζεται με το πώς μπορούμε να κάνουμε τις πόλεις ελκυστικές για την επιχειρηματικότητα. Πώς θα μπορέσουν οι πόλεις, τα αστικά κέντρα να είναι χώροι δημιουργίας ευκαιρίας για να ξεκινήσουν νέες επιχειρήσεις, για να αναπτυχθούν είτε ώστε μεγάλες πολυεθνικές π.χ. επιχειρήσεις να αποφασίζουν να εγκατασταθούν εκεί. Μεταξύ των διαφόρων έργων και προγραμμάτων που έχετε στην γύρωσή της έχετε και μια εξαιρετική ιστοσελίδα όπου βρίσκει κανείς πολλές πληροφορίες. Έχετε φόρουμ, έχετε ομάδες εργασίας και βλέπω πάρα πολλές πρωτοβουλίες για την υποστήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ή για, την, για τα προγράμματα κατάρτισης, αλλά δεν έχω δει συγκεκριμένα έργα, τουλάχιστον όχι στην ιστοσελίδα, ή τουλάχιστον δεν τα βρήκα εγώ, για την ανάπτυξη, την οικονομική ανάπτυξη δηλαδή των πόλεων, γιατί προκειμένου να είναι οι πόλεις ε, ε, επαρκής ικανοποιητική χώρη για τη ζωή των πολιτών πρέπει να έχουν μια πλούσια οικονομική δραστηριότητα. Επίσης ήθελα να σας ρωτήσω ε, ποιος είναι ο λογισμός του γύρω της με, με, τι πόρους κινείστε για όλα αυτά τα προγράμματα και τις ε, πρωτοβουλίες που βλέπουμε. Σας ευχαριστώ κύριο Σαϊμό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έρχομαι από το Ανατολικό Βέλγιο, στην οριακή περιοχή. Είμαι πολύ κοντά σε τρία σε σύνορα τριών χωρών. Είμαι και εγώ λοιπόν πεπισμένο Ευρωπαίο όπω και ο παππού σα. Όταν ήταν υπουργό, ε, επίτροπο εδώ, τότε εγώ ήμουν βοηθό. Ε, και ο παππού σα ε, ήταν ένα μεγάλο Ευρωπαίο και Ευρωπαϊστή. Είστε δήμαρχο μια από τι πιο όμορφε πόλει τη Ευρώπη. Αυτό είναι... Ε, αυτό που σα λέω είναι αλήθεια. Ο δεν έχει πάει στη Γάντη πρέπει να πάει είπατε στην ομιλία σας ότι η πόλη είναι ένας σημαντικός εταίρος, απαραίτητος και έχετε απόλυτο δίκιο. Και αυτό που θα μας παρουσιάσει την ερχόμενη εβδομάδα κυρία Φόντε με το Green Deal, το Ευρωπαϊκό Green Deal θα εφαρμοστεί κυρίως στις πόλεις διότι εκεί ζουν και περισσότεροι άνθρωποι. Υπάρχουν ζητήματα συνύπαρξης, ε, μεταφορών, ε, ζητήματα ενεργειακά. Για να επιλύσουν τα ζητήματα αυτά, οι λύσει είναι στην πόλη. Επίσης είπατε ότι πρέπει να είναι πιο ισχυρή η πολιτική συνοχής. Το είπε και ο πρόεδρος. Είμαι εισηγητής ε, για το Interreg και πρέπει να πω ότι διαπιστώνω ότι η αρχική των κυβερνήσεων, το Συμβούλιο έχουν υποβάλει μια νέα πρόταση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο όπου αυτό τόσο μικρό πρόγραμμα, το Interreg, θα μειωθεί η χρηματοδότηση 30%. Υπάρχουν άνθρωποι που εφαρμόζουν αυτό το πρόγραμμα και αυτοί οι άνθρωποι είναι που έχουν την Ευρώπη στην καρδιά τους. Και αυτοί οι άνθρωποι διαμαρτύρονται. Λένε ότι το πρόγραμμα αυτό θα εκλείψει εσείς ε, ως ε, μέλος της EuroCity πώς μπορείτε να πείσετε ε, ότι τους αρχηγούς των κυβερνήσεων δεν πρέπει να λάβουν χώρα αυτές τις περικοπές. Δεύτερον. Για τα παιδιά είναι καταπληκτικά, αλλά θα ήθελα να σας δώσω ήθελα να εκφράσω μια ε, επιθυμία για τον, Άγιο Νικό, για τον Άι Βασίλη. Ποια θα ήταν η ευχή σας προς τον Άι Βασίλη την 1η Ιανουαρίου του 2020 η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και ειδικότερα όσον αφορά τα περιφερειακά ταμεία να αλλάξει ούτω ώστε οι πόλεις να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν, ποιο ένα μέτρο θα, ε, στέλνατε, θα κάνατε ως ευχή στον Άγιο Βασίλη εσείς ως Δήμαρχος. Merci beaucoup, Pascal. Euh, Julie Ward. Η Judy Ward έχει το λόγο, παρακαλώ. Uh, thank you very much. Uh, I've also uh, made the journey from Brussels to... Ναι, και εγώ έχω πάει στη Γάνδη. Ε, δεν έχω καταφέρει βεβαίως ε, να δω το Βέλγιο όσο θα ήθελα από τότε που έχω εκλεγεί, αλλά είδα εκεί στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης ε, φοιτητές, καθηγητές, ε, που ασχολούνται με καλλιτεχνικές σπουδέ. θα ήθελα να αναφερθώ και στην σημασία του πολιτισμού στις πόλεις. Ε, πώς αντιλαμβάνεστε εσείς τη σημασία του. Είναι ένας φορέας οικονομικής αναζωγόνησης. Πώς όμως εσείς βλέπετε το θέμα αυτό της ε, gentrification, όπου δηλαδή έρχονται καλλιτέχνες ε, και ε, καταλαμβάνουν περιοχές ολόκληρες. Ε, Βεβαίω, αυτέ οι περιοχέ ξαφνικά γίνονται ενδιαφέρουσε, γίνονται πολύ πιο όμορφε, αλλά κάποιοι άνθρωποι που ζούσαν εκεί δεν μπορούν πια να ζήσουν εκεί γιατί ανεβαίνουν οι τιμέ. Εγώ προέρχομαι από τον τομέα αυτών τη δημιουργία και νομίζω ότι πρέπει πραγματικά να προσέξουμε τους καλλιτέχνες μας, την κοινότητά μας των καλλιτεχνών, όχι μόνο επειδή μας δίνουν τη δυνατότητα, δίνουν τη δυνατότητα στις πόλεις να μεγαλώνουν και να ζωγονώνται. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, ο λογικό τομέα ήταν πιο ανθεκτικούς και εκπροσωπούν πολύ μεγαλύτερο μέρος του ΑΕΠ από ότι κάποιες άλλες παραδοσιακές μορφές ε, δραστηριοτήτων. Πώς λοιπόν μπορεί, θεωρείτε εσείς, ότι ο τομέας της δημιουργίας μπορεί να αντιμετωπίσει και κάποιες εντάσεις που υπάρχουν στις κοινωνίες μας. Ε, υπάρχουν σημαντικά θέματα, έτσι. Ε, ο φόβος του άλλου. Ε, στις πόλεις έρχονται καινούργιοι άνθρωποι συνεχώς, πρόσφυγες, μετανάστες, συνήθως πάνε στις πόλεις. Στην πόλη μου, το Μάντσεστερ, υπάρχει, έχει δημιουργηθεί μια ε, πολύ σπουδαία δυνατότητα ε, να ζουν μαζί άνθρωποι από διαφορετικούς ορίζοντες και ο πολιτισμός ε, είναι ο τόπος για να συναντηθούν αυτές οι κουλτούρες, να γίνει αυτός ο διάλογος. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορέσαμε να οθήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε ο πολιτισμός και η εκπαίδευση να επιστρέψουν ε, στην, το χρωτοφυλάκιο της κυρίας Μαρία Γκαμπριέλ. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Όμω, στα πλαίσια του Eurocities που συζητούμε σήμερα, ξέρω ότι ο, πολ, πολιτισμό ε, ε, και εκεί λαμβάνει την υπόψη. Θα ήθελα να ξέρω πόσο εσεί το προωθείτε το θέμα του πολιτισμού και κατά πόσο αυτό μπορεί να βοηθήσει και την πράσινη ατζέντα, το Green Deal διαπιστώσατε ότι ε, η παρέμβασή σας ε, οδήγησε σε πολλά σχόλια, πολλές παρατηρήσεις και είμαστε στη διάθεσή σας ε, για να ακούσουμε τις απαντήσεις σας. δεν ήμουν βεβαίω στο κοινοβούλιο την ίδια εποχή που ανέφερε και εσύ, αλλά είναι αλήθεια ότι ο παππούς ήταν σπουδαίος ευρωβουλευτής, άφησε, ε, ο σπουδαίος επίτροπος ε, άφησε το σημάδι του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με αυτά που είπατε και με αυτά που έχετε κάνει είστε και εσείς ένας σπουδαίος Ευρωπαίος και όλοι είμαστε με κάποιο τρόπο με τις αξίες που φέρουμε εδώ στην Επιτροπή Ρέτζι. Η Επιτροπή Ρέτζι είναι πολιτικά ποικιλόμορφη βέβαια, αλλά υπάρχουν σειρά από που μας ενώνουν. Αυτή είναι και η ισχύς μας. Λοιπόν, σας δίνω τη δυνατότητα να απαντήσετε και στους δύο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Πραγματικά νιώθω ότι θα είστε ένας εταίρος στην προσπάθειά μας έτσι ώστε οι περιφέρειες και ιδιαίτερα οι πόλεις να βγουν στην ατζέντα των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και θέλω να σας ευχαριστήσω ε, για αυτήν την υποστήριξη. Να πω κάποια πράγματα, θα δώσω βεβαίως και το λόγο στην Γενική Διευθύντρια, την Αναλύσα Μπονή. Ε, πρώτα απ' όλα να ε, αρχίσω από εκεί που τελείωσαν οι παρεμβάσεις για το Manchester. Ο Κέβιν De Bruyne, ε, ξέρετε, παίκτη τη Manchester City, είναι από τη Γάνδη. Είναι από του καλύτερου του κόσμου. Είναι από την πόλη μου. Οι γονεί του ζουν 5 χιλιόμετρα από το σπίτι μου. Και παίζει στο Manchester ποδόσφαιρο. Ή έπρεπε να το πω και αυτό. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε για τον πολιτισμό και του καλλιτέχνε. Στην πόλη τη Γάνδη, εμείς έχουμε ένα προπολογισμό για τον επόμενα πέντε έτη και τετραπλασιάσαμε τον προπολογισμό για τις πολιτιστικές υποδομές. Διότι είμαστε πεπισμένοι ότι η ανανέωση πολιτιστική είναι και η βάση για την οικονομική ανάπτυξη στις πόλεις μας. Δεν είναι θέμα το να επιλέξουμε είτε πολιτισμός είτε επιχειρήσεις. Όχι, αυτά είναι πράγματα τα οποία πάνε μαζί. Ε, κύριε Μότεκ, μιλήσατε για τα ζητήματα στέγασης. Εμείς θέλουμε να είναι προσβάσιμοι, προσβάσιμες κατοικίες με τον δήμαρχο της Πράγας, ε, της Φλωρεντίας, ε, ε, της Βαρσοβίας, ο Ντάριο Ναρντέλα, ο, δήμαρχος της ε, ε, Φλωρεντίας 42 χρονών, 38% μέχρι της Πράγας, 37 χρονών εγώ. έχουμε μια νέα γενιά δημάρχων κατά κάποιο τρόπο σε τοπικό επίπεδο, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο. Και αυτό είναι καλό. Ήθελα να πω εδώ στην Ισπανίδα κυρία ότι η ελκυστικότητα για τις επιχειρήσεις αν θέλουν δηλαδή να επενδύσουν στην πόλη μου παραδείγματος χάρη το πρώτο ερώτημα πάντα είναι κατά πόσο υπάρχουν δημόσιες, μετα, δημόσιες μεταφορές, ε, κατά πόσο ε, δεν υπάρχει συμφόρηση. Πάνε χέρι-χέρι αυτά και αυτό είναι στα χέρια ε, της τοπικής πολιτικής. Δεν είναι οι μεγάλες ιδεολογικές συζητήσεις. Οι πράσινοι, οι σοσιαλιστές λένε να μην υπάρχουν αυτοκίνητα. Ε, όχι, ακούστε, εγώ είμαι φιλελεύθερος, ε, αλλά είμαι πεπισμένος ότι χρειαζόμαστε και δημόσιες μεταφορές και να μην υπάρχει συμφόρηση. Ιδάλλως οι επιχειρήσεις δεν θα επενδύσουν στην πόλη μας. Στην πόλη μας, πριν από 10 χρόνια σε 10 χρόνια ελπίζουμε να έχουμε 10.000 νέες θέσεις εργασίας γιατί έχουμε επενδύσει και έχουμε φιλοδοξία στον τομέα των μεταφορών, στον τομέα των υποδομών. Οι μεγάλες δελογικές συζητήσεις ε, ορισμένε φορές ε, σε εθνικό επίπεδο ε, μιλάμε πολύ αλλά δεν παίρνουν τα αποφάσεις. Σε τοπικό όμως επίπεδο εμεί αποφασίζουμε και το κάνουμε μαζί όλα τα πολιτικά κόμματα για να προχωρήσουμε για την πόλη μας, να κάνουμε δουλειά πάνω σε αισθήματα στέγασης, σε αισθήματα κινητικότητας. Δεν μπορούμε να έχουμε μια μεγάλη ευημερούσα πόλη αν δεν μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση στην κατοικία. Έχουμε μεγάλα λιμάνια, ξέρετε η Κοπεχάγη και το Μάλμοε ε, έχουν αυτό το μεγάλο ε, ε, μεγάλη γέφυρα. Η δεύτερη μεγαλύτερη γέφυρα είναι η δικιά μας από τη Ζέλαντ στην Ολλανδία εδώ στη Γάνδη. αλλά πρέπει και οι άνθρωποι που εργάζονται να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην κατοικία, να έχουν εκπαίδευση για τα παιδιά τους. σε τοπικό επίπεδο λοιπόν, χωρίς να μπαίνουμε σε μεγάλα ιδεολογικά ζητήματα, ρεαλιστικά ε, προχωράμε ρεαλιστικά και ενωμένα. Η αναλύση θα σας πει ότι εμείς ε, θέλουμε πραγματικά να ενθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις να έρθουν να επενδύσουν σε εμά. Τώρα, η ευχή μας είναι να, αυτό που θέλουμε μάλλον εμείς είναι να έχουμε και εμείς ως πόλεις ε, λόγο Θέλουμε να είμαστε στο τραπέζι όπου παίρνονται οι αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γνωρίζω πολύ καλά τον Σαρλ Μισελ, ήταν ο πρώην πρωθυπουργό μας. Εμείς έχουμε μια ευθύνη ως επικεφαλής κάποιων πόλεων να μπορούμε να πούμε στους διάφορους αρχηγούς κρατών, στα θεσμικά όργανα, αγκαλιάστε τις πόλεις, ελάτε να συζητήσουμε, ελάτε να πραγματοποιήσουμε από κοινού τις φιλοδοξίες μας. Έχει ο καθένας φιλοδοξίες το Συμβούλιο, η Κομισιόν, αλλά αυτοί οι στόχοι θα επιτευχθούν μόνο με τις πόλεις. Μόνο εφόσον οι πόλεις έχουν και αυτές λόγο. Είναι μια συγκεκριμένη πρόταση λοιπόν αυτή. Δεν θέλουμε να δημιουργηθεί κάποια νέα οργάνωση, κάποιο νέο φόρουμ ή να γίνει κάποια διάσκεψη. Θέλουμε οι πόλεις να είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορούμε ε, να πείσουμε μέσω της συζήτησης τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, να έχουμε λοιπόν λόγο. Διότι έρχονται έτσι οι πολίτες και πιο κοντά στις ευρωπαϊκές πολιτικές όταν βλέπουν ότι έχουν λόγο στη διαμόρφωσή τους. Τώρα για την πολιτική συνοχής ε, ε φτωχές περιοχές, όλες τις περιοχές. Εμείς πιστεύουμε ότι, ότι όλες τις περιοχές, όλες οι περιφέρειες πρέπει να έχουν μια πολιτική συνοχής. Δεν ξέρω αν η Αλίσσα θέλει να προσθέσει κάποια πράγματα. Ευχαριστώ ξανά εκ τη της ε, Σίτη. Ε, ευχαριστούμε για αυτή την πολύ δραστήρια συμμετοχή και για τι ερωτήσει σα. Καιρό ε, ασχολούμαι με το Σίτη και ποτέ δεν είχα τόσο ωραίε αντιδράσει. Είναι πολύ καλό αυτό. Σα ευχαριστώ. Λοιπόν, όσον αφορά τι διαφορέ ερωτήσει τώρα, για τα όσα είπατε για την πολιτική συνοχή. φυσικά θέλουμε μια ανοιχτή πολιτική συνοχή προ όλε τι περιφέρειες. Κυρίω επειδή παρατηρούμε ότι πολλές από τις προκλήσεις, τουλάχιστον όπω το βλέπουμε εμεί είναι ίδιες παντού ε, στην Ευρώπη. Ε, το ζήτημα του κλίματος είναι ένα πρόβλημα παντού. Το πρόβλημα της φτώχειας, ε, ειδικά τώρα στις μεγαλοπόλεις, ισχύει για όλες τις μεγαλοπόλεις. Οι φθηνές κατοικίες, οι κατοικίες, η καινοτομία, όλα αυτά είναι θέματα που υπάρχουν παντού. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μην κάνουμε διαχωρισμούς μεταξύ Ανατολικής Ευρώπης, Δυτικής Ευρώπης, νέων χωρών. Είναι σημαντικό η πολιτική συνοχή να παραμένει ε, ε, να παραμείνει σαν ένα συνδετικό υλικό, σαν μια κόλλα για όλη την Ευρώπη και ισχυρή όσον αφορά τον προϋπολογισμό και το όραμα για να ενισχύσει την Ευρώπη. Ε, θα πρέπει να παραμείνει έτσι για όλους. Uh, το ζήτημα που αναφέρατε και ο Ρικάρντο Ρίο είναι ένας από τους καλύτερους ε, δημάρχους μας. Είναι δραστήριος, έχει μεταμορφώσει την πόλη του με καταπληκτικό τρόπο μέσα σε λίγα χρόνια στην Πορτογαλία. Αυτή η ιδέα της συνεργασίας, το να μην δημιουργεί ε, αστικές συγκρούσεις, είναι πραγματικά χαζό το να μιλάμε, πρέπει να μιλάμε για αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν. Στη δουλειά μας αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να προσπαθούμε να επισημαίνουμε τη σημασία των μεγαλοπόλεων, των μεγάλων αστικών κέντρων. Διότι αυτή η συνεργασία όλων των Δήμων ε, σε έναν μεγάλο χώρο που δεν είναι απόλυτα αστικός αλλά είναι λειτουργικός είναι ένας τρόπος ε, ε, να συνδεθούμε και με τις πιο αγροτικές περιοχές με όλες τις σχετικές ε, υπηρεσίες και λειτουργικότητες που χρειάζεται η περιοχή αυτή Και φυσικά και οι μεταφορέ είναι πάρα πολύ σημαντικέ, οι συγκοινωνίε, αλλά και η δημιουργία θέσεων εργασία, ε, η αγορά εργασία και ούτω καθεξή. Είναι κάτι που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε κάποιο είδου ε, δεσμού αντί να γεννάμε διαφορέ. Ειδικότερα όσον αφορά το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Και εκεί δεν πρέπει να έχουμε τέτοιο διαχωρισμό να μην ε, χωρίζουμε τα συμφέροντά μα. Πρέπει να βρούμε τρόπου να συνδεθούμε παραπάνω, να δούμε πόσο ω θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε καλύτερα ε, και με τα αγροτικά λόμπι για να βρούμε νέου τρόπου. Η ελκυστικότητα των πόλεων και ούτω καθεξής. Ε, επίσης οριζόντιο ζήτημα που αφορά πολλούς τομείς. Ε, προτεραιότητα για τις πόλεις αφορά την ανανέωση, το χρήση του χώρου, τη χωροταξία, ε, την προβολή των πόλεων, την επιχειρηματικότητα με πάρα πολλούς τομείς. Έχουμε πολλές διαφορετικές ομάδες εργασίας που ασχολούνται με αυτό. Φυσικά η οργάνωσή μας, η οποία παρεμπιπτόντως ε, έχει ένα προϋπολογισμό περίπου 4 εκατομμυρίων και χρηματοδοτείται κυρίως από τις συμμετοχές των μελών, αλλά έχουμε και κάποια προγράμματα, κάποια έργα τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία μας επιτρέπουν να εμβαθύνουμε σε κάποιους τομείς. Το δίκτυό μας λοιπόν είναι οργανωμένο γύρω από κοινότητες. Ανθρώπους που προέρχονται από δημοτικ τις διοικήσεις ε, και υπάρχει μια οργάνωση τομεακή γιατί όλες οι διοικήσεις όπως και το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν όλα τα επίπεδα διοίκησης δεν πάβουν να είναι οργανωμένα να τομίσει ο πολιτισμός, η οικονομική ανάπτυξη, η ε, ψηφιακή διάσταση, το περιβάλλον, οι μεταφορές και το καθεξής. Αλλά φυσικά όλο και περισσότερο και θα το έχετε παρατηρήσει στη δική μας περιγραφή του στρατηγικού μας πλαισίου υπάρχουν μεγάλες ανάγκες συνεργασίας διακλαδικής και πιο ολοκληρωμένη γιατί η πραγματικότητα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι πολύ πιο περιπλοκή από απλά περιβάλλον ή απλά μεταφορέ. Εφαρμόζουμε λοιπόν αυτό τον τρόπο εργασία και αυτό θα επηρεάσει και το πώ θα προβούμε στο να επιτύχουμε την ε, βελτίωση τη ελκυστικότητα των πόλεων, την αναγέννηση των πόλεων. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να συνεργαστούμε πιο συγκεκριμένα για αυτές τις πτυχές. Για τον πολιτισμό απαντήσατε. Για το πράσινο σύμφωνο, για το Green Deal, που δεν είναι πια τόσο νέο. Το Ευρωπαϊκό Πράσινο Σύμφωνο. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτό το επίπεδο. Ο Αντιπρόεδρος Τίμερμανς θα χρειαστεί, πιστεύουμε, να συνεργαστεί με τις πόλεις. Διότι υπάρχουν φιλοδοξίες και γιατί τελικά οι ίδιοι οι πολίτες θα κάνουν την αλλαγή. Αυτοί θα αλλάξουν τα πράγματα όσον αφορά το κλίμα. Αυτοί θα αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους, τον τρόπο κατανάλωσής τους και οι δημοτικές αρχές με τις κατάλληλες φιλοδοξίες θα μπορέσουν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις, αλλά οι πολίτες είναι εκείνοι οι οποίοι θα χρησιμοποιούν τις συγκοινωνίες, θα καταναλώνουν λιγότερα και όλα αυτά. Εκεί λοιπόν πιστεύω ότι οι πόλεις μπορούν να βοηθήσουν να υλοποιήσουμε αυτό το βουνό που μας περιμένει από υποχρεώσεις. Και πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, ότι οι Κομισιόν και το Κοινοβούλιο μπορούν να βασιστούν σε εμά. Θα προτείνουμε λύσει, ε, ε, τεχνογνωσία για να δούμε πώ μπορούμε να ανακαινήσουμε όλα αυτά τα κτίρια ε, τα οποία θα παίξουν σημαντικότατο ρόλο για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Τι είδου συστήματα δηλαδή μπορούμε να συμπεριλάβουμε στο Πράσινο Σύμφωνο που θα μπορούσαν να εφαρμόσουν οι πόλει, οι Δήμοι σε όλους τους τομείς. Ε, έχει ανοίξει λοιπόν ο διάβλος επικοινωνίας. Θα πρέπει να καθίσουμε όλοι μαζί στο τραπέζι ε, όπου χαράσεται η ευρωπαϊκή πολιτική. Αν μπορούσαμε εμείς να συμμετέχουμε στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση πολιτικών που παίζουν σημαντικό ρόλο για τις πόλεις, θα μπορούσαμε να φέρουμε καλύτερα αποτελέσματα στην εφαρμογή διότι έτσι θα τις υιοθετήσουν πιο εύκολα οι άνθρωποι, θα τις δεχτούν πιο εύκολα οι άνθρωποι και θα μπορούμε να τις υλοποιήσουμε καλύτερα ε, στην πραγματικότητα. Είναι μια κατάσταση με την οποία κερδίζουν όλοι, αλλά ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί έτσι που δεν επιτρέπει επίσημα στις πόλεις να συμμετέχουν ε, σε αυτές τις συζητήσεις, εντάξει μόνο στην Επιτροπή των Περιφερειών βέβαια, αλλά φυσικά όπως έχουμε πει πολλές φορές είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με την Επιτροπή σας αλλά και με άλλες επιτροπές, δίνοντας σας ιδέες, υποστήριξη. Θεωρήστε μας ε, στρατηγικούς εταίρους για την υλοποίηση των δικών σας προγραμμάτων. Οι Ιταλικές πόλεις ελπίζω το σημείωσα. Να μπορείτε να μας βοηθήσετε, κύριε Ντονάτο. Θα ήθελα να μάθω παραπάνω, κύριε Ντονάτο, γι' αυτό. Νομίζω τα καλύψαμε όλα. Ευχαριστούμε, Αναλίζα. Εγώ ήθελα να σας πω ότι δεν έχω επισκεφθεί την ε, Γανδί, είναι κενό από πλευράς μου. Πέρα από τα ιστορικά και του Ερίκου του Πέμπτου, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να πάω γιατί βλέπω ένα δήμαρχο με όραμα, με ενθουσιασμό και εμείς ε, που είμαστε που έχουμε διαγράψει μια πολιτική σταδιοδρομία όταν ακούμε έναν νεαρό δήμαρχο σαν και εσάς έχουμε περισσότερη πίστη και ελπίδα για το μέλλον. Και γι' αυτό θέλω να έρθω στην πόλη σας βρισκόμαστε σε μια στιγμή όπου πραγματικά σας χρειαζόμαστε. Έχουμε μπροστά μας διαπραγματεύσεις ε, ε, διοργανικές, θεσμικές, για να διασώσουμε μια φιλόδοξη πολιτική περιφερειακή και έναν φιλόδοξο προϋπολογισμό. Γιατί το ένα δεν μπορεί να γίνει χωρίς το άλλο. Αλλά στην πραγματικότητα Χρειαζόμαστε στήριξη. Στήριξη που θα φέρνουν στο προσκήνιο το έδαφος, την περιφέρεια της πόλης με όλα τα επιχειρήματα που μας αναφέρατε, τις προκλήσεις, την κλιματική αλλαγή, την ε, ένταξη των μεταναστών, τα δίκτυα των μεταφορών θα μπορέσουν να επιληθούν αυτά μόνο αν έχουμε τα μέσα, τους πόρους, διάθεσή μας. Και γι' αυτό είναι σημαντικό και είχα προτείνει αυτό το θέμα και την συζήτηση με τη EuroCities να οργανωθούν οι πόλεις, οι δήμαρχοι, οι δήμοι, να επεξεργαστούν ενδεχομένως και μια διακήρυξη σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να την αποστείλουμε στο Συμβούλιο ότι έχουμε φτάσει στο όριο και να για ποιους λόγους σχετικά με, τους, ε, με τις προτάσεις προϋπολογισμού σας για τη μελλοντική πολιτική. Εάν συνδυαστούν δήμοι μεγάλων και μικρότερων πόλεων από τη Γάνδη, από τη Λισαβόνα, από το Παρίσι και λέει ο πρόεδρος, αυτό θα έχει πολιτική ισχύ. Και εμείς θα το βλέπαμε ως βοήθεια, ενίσχυση στο δύσκολο έργο και διαπραγμάτευση που έχουμε μπροστά μας. Είμαστε λοιπόν στη διάθεσή σας για να οργανώσουμε κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε μεγάλα χρονικά περιθώρια. και έχουμε πολιτικές στοχεύσεις που απαιτούν από εμά να είμαστε παρόντες. Είμαι σίγουρος ότι συμφωνούν οι συνάδελφοι ε, εκφράζοντας την ικανοποίησή μας για την ανταλλαγή αυτή που είχαμε σήμερα που δεν ήταν σίγουρα η τελευταία αλλά ήταν ο πρώτος φορέας δίκτυο που θα έλαμε εδώ να καλωσορίσουμε στην Επιτροπή. Ευχαριστούμε λοιπόν. Συνεχίζουμε λοιπόν με την ε, ημερήσια διάταξη με θέμα εξίσου σημαντικό και που αφορά την παρουσίαση του κυρίου Σπάιχ που με χαρά υποδέχομαι ο οποίος επεξεργάστηκε όπως τα γνωρίζετε την έκθεση για την Επιτροπή των Περιφερειών που θα έχετε ελπίζω διαβάσει όλοι για τις περιφέρειες του Άνθρακα. Είναι ένα θέμα επίκαιρο και πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω σήμερα ή εχθές άνοιξε το συνέδριο για το κλίμα στη Μαδρίτη, η διάσκεψη και έχουμε και τον κανονισμό της Επιτροπής για το Ταμείο της Δίκαιης Μετάβασης όπου έχουμε τον ρόλο του συνομοθέτη να διαδραματίσουμε, χρειαζόμαστε πληροφορίες, ενημέρωση και νομίζω ότι η συνεισφορά της Επιτροπής των Περιφερειών είναι πολύ ενδιαφέρουσα, θα μας επιτρέψει να λάβουμε τις καλύτερες ε, αποφάσεις που μπορούμε. Έχετε λοιπόν το λόγο για 15 με 20 λεπτά, λέει ο Πρόεδρος, για να κάνουμε συζήτηση μετά με τους συναδέλφους. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σήμερα. Αξιότιμε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέλη της Επιτροπής Ρέτζη, κυρίες και κύριοι, είμαι εξαιρετικά ευγνώμων που έχω τη δυνατότητα να μιλήσω εδώ ενώπιον της Επιτροπής αυτής, διότι αυτό δείχνει την πόσο καλή σχέση έχουμε ε, αφενός δηλαδή η Επιτροπή των Περιφερειών και αφετέρου η Επιτροπή Ρέτζη. Ο πρόεδρος μας, ο κύριος ε, Λάμπερτς, είχε τη δυνατότητα να συζητήσει μαζί σας ε, τις εργασίες του στην Επιτροπή των Περιφερειών. Είχαμε και μια κοινή συνάντηση με την Επιτροπή για την Εδαφική Συνοχή, για τον προϋπολογισμό και χαίρομαι βέβαια που και εσείς προσωπικά κύριε Πρόεδρε ήρθατε σε ένα πάνελ που οργάνωσε η Επιτροπή Περιφερειών ε, για την μετάβαση, την κοινωνικονομική αλλαγή περιπτώσει, στι περιοχέ παραγωγή άνθρακα είναι κάτι που είναι απαραίτητο αν θέλουμε να κινηθούμε προ αυτή την κατεύθυνση. Είναι τεράστιε όμω και οι προκλήσει που συνδέονται με αυτήν την ανάγκη αφενός αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, αφετέρου ε, να μπορέσει αυτή η αλλαγή να γίνει κοινωνικώς αποδεκτή. Αυτό είναι και, ε, αυτός είναι και ο πυρήνας της νομοδότησής μου στην Επιτροπή των Περιφερειών. Πρέπει να εξηγήσω ότι αυτό είναι κάτι που συνδέεται και ε, με τον περιβάλλον από που προέρχομαι. Προέρχομαι από τη Βόρεια Βεσταλία στη Γερμανία, έχω εργαστεί στα ζητήματα αυτά. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ομοσπονδοκρατήδιο με 18 εκατομμύρια κατοίκους είναι και η καρδιά της γερμανικής βιομηχανοποίησης ήταν πάντα η καρδιά της γερμανικής βιομηχανίας ε, ήδη από το 19ο αιώνα. Αυτή η διαδικασία βεβαίως βασίστηκε κυρίως στον άνθρακα και στο χάλιβα. Ήταν ε, ουσιαστικά η βάση του ε, γερμανικού οικονομικού θαύματος. Αυτός ο χάλιβας όμως που ε, έφερε την εφημερία χρησιμοποιήθηκε και για να εξοπλίσουμε το στρατό μας που έφερε αυτούς τους δύο φοβερούς πολέμους στην Ευρώπη. Ε, έτσι λοιπόν βλέπετε ότι ο Χάλιβας μπορεί να φέρει ευημερία, μπορεί να φέρει και καταστροφή. Αυτά βεβαίω οδήγησαν και ο Χάλιβας επίσης οδήγησε στη δημιουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την ε, Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα. Πέρσι κλείσαμε ε, το τελευταίο ορυχείο μετά από 200 χρόνια. Το τελευταίο ορυχείο άνθρακα. Κάποτε εργαζόντουσαν 500.000 άνθρωποι στον τομέα αυτόν. Και τώρα δεν είναι κανείς. Ήταν μια επίπονη διαδικασία όπως αντιλαμβάνεστε, όμως αυτή η διαδικασία ε, είχε να κάνει με την έλλειψη ανταγωνιστικότητας δεν είχε πλέον νόημα, δεν ήταν ανταγωνιστικό να κατεβαίνουμε 1200 μέτρα μέσα στη γη όταν μπορεί κανείς να εισάγει άνθρακα από την Αυστραλία, από αλλού, με, λιγότερα χρήματα. Βεβαίως, δύο είναι τα διδάγματα από τη διαδικασία αυτή. Το πρώτο είναι ότι όταν περνάμε σε μια τόσο σημαντική αλλαγή, ε, χρωστάμε κάτι στους εργαζόμενους αυτού του κλάδου. Στους ανθρώπους οι οποίοι διακύβευσαν την υγεία τους, τη ζωή τους ορισμένες φορές για να μπορέσουν να προσφέρουν την ενέργεια την οποία χρειαζόντουσαν βιομηχανίες ε, και βεβαίως χρειάστηκαν και πολλά χρήματα για να γίνει κοινωνικώς αποδεκτή αυτή η μετάβαση. Ε, θα θυμάστε τις εικόνες ε, με τους αστυνομικούς ε, ε, που πάνω σε άλογα ε, που χτυπούν ε, διαδεδοτές ανθρακορίχους. Αυτά δεν έγιναν σε εμά. Δεν έγιναν στη δική μας περιφέρεια. Βεβαίως δεν επενδύσαμε επαρκώς στο μέλλον προς νέες αλυσίδες αξιών, προς νέες νέους τομείς δημιουργίας τη απασχόλησης. Αυτό είναι ένα κεντρικό δίδαγμα που θέλουμε ε, να μεταφέρουμε σε αυτή τη διαδικασία τη μεταβατική. Βεβαίως τώρα το σημείο αφιτερίας είναι πολύ διαφορετικό. Δεν μιλάμε πλέον για έλλειμμα ανταγωνιστικότητας. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια πολιτική απόφαση. Η πολιτική απόφαση να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Η Συμφωνία των Παρισίων είναι η βάση αυτή της διαδικασία μετάλλαξη. Και είναι σωστή αυτή η απόφαση. Έπρεπε να πάρουμε αυτή την απόφαση, την θαραλέα και έπρεπε να σταματήσει η παραγωγή άνθρακα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Διότι ο άνθρακα είναι στην καρδιά του προβλήματο που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Αυτή λοιπόν η διαδικασία μετατροπή είναι πολιτικώ απαραίτητη. Αυτό που θέλω να καταστήσει Βεβαίω από την άλλη είναι και μια πολιτική απόφαση η οποία έχει τεράστιο αντίκτυπο στους ανθρώπους που ζουν στις περιοχές αυτές ε, ε, παραγωγής άνθρακα. Και οι θέσεις εργασίας που συνδέονται με την παραγωγή άνθρακα είναι καλοπληρωμένες και είναι οι μόνες καλοπληρωμένες ε, θέσεις εργασίας αυτές τις περιοχές ορισμένες φορές. Χρειαζόμαστε λοιπόν πραγματικά, πραγματικά ανταγωνιστικές ε, αλυσίδες αξιών ε, σε αυτές τις περιοχές. Πρέπει να βρούμε λύσεις για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που εργάζονται στον άνθρακα έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις αυτές και να τους δώσουμε νέες προοπτικές. Αυτό ήταν και στην καρδιά της νομοδότησής μου στην Επιτροπή των Περιφερειών. Και βέβαια στο σημείο αφετηρίας είναι ε, τα υπάρχοντα εργαλεία αρκούν για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την τεράστια ε, διαδικασία μετατροπής. Και πολύ γρήγορα η συζήτηση ε, έφτασε και στο Ταμείο Δίκαιης ε, Μετάβασης, κάτι που προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βέβαια, και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό, χρειαζόμαστε αυτό το εργαλείο για να μπορέσει να λάβει η χώρα αυτή η τόσο σημαντική αλλαγή τα πιο πρόσφατα σχόλια του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής, της της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, έλαβαν υπόψη αυτό το γεγονός και χαίρομαι γι' αυτό. Ε, θέλω εδώ να υπογραμμίσω τρία σημεία κλειδιά. Πρώτα απ' όλα είμαι πεπισμένος ότι πρέπει αυτά τα χρήματα να είναι επιπλέον χρήματα. Αν προέλθουν από τα ταμεία συνοχής ε, τα χρήματα αυτά, τότε η λογική πια θα είναι περίεργη αφαιρούμε χρήματα από φτωχέ περιοχές για να, για βοηθήσουμε περιοχές που μπορεί να ε, φτωχύνουν στο μέλλον. Ε, δεν είναι λογικό αυτό. Χρειάζονται καινούργια χρήματα. Δεν πρέπει να ε, φέρουμε σε αντιπαράθεση τις, τις διάφορες περιφέρειες της Ευρώπης μεταξύ τους. Το δεύτερο σημείο κλειδί. Αυτό το οικονομικό μέσο, αυτό το ταμείο θα πρέπει να συνδέεται με την περιφερειακή πολιτική γνωρίζω ότι στην αρχική πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπήρχε αυτή η ιδέα ενός ταμείου το οποίο θα διαχειριζόμαστε κεντρικά στις Βρυξέλλες. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι σωστό. Και το λέω αυτό εδώ στην Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής. Χρειαζόμαστε ε, προσεγγίσεις που να προσαρμόζονται στην κάθε περιοχή. Είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Είναι διαφορετικά τα προαπαιτούμενα. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Χρειαζόμαστε λοιπόν προσεγγίσει ε, προσαρμοσμένε. Ε, όπου θα βασιζόμαστε στη γνώση των συντημάτων της κάθε περιοχής. Υπάρχει αυτή η αρχή ε, της ε, συνευθύνης ε, στην πολιτική συνοχή, η οποία είναι απαραίτητη και εδώ. Πρέπει λοιπόν να συνδέσουμε αυτή την προσπάθεια με την πολιτική συνοχή και δεν θέλουμε να διαχειρίζονται, να διαχειρίζονται όλα αυτά εδώ στις Βρυξέλλες κεντρικά. Ε, και τώρα θα ήθελα να μιλήσω για τις κρατικές ενισχύσεις και τη σχετική πολιτική. Θα πρέπει πραγματικά να σκεφτούμε εκ νέου τα διάφορα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Η υπάρχουσα οικονομική κατάσταση είναι το πιο σημαντικό. Εδώ όμως αυτό που θέλουμε εμείς είναι να αποφύγουμε οι περιοχές οι οποίες επηρεάζονται από αυτές τις αλλαγές να φτωχύνουν στο μέλλον. Δηλαδή πρέπει να επενδύσουμε τώρα για να μην υπάρξει επιδείνωση της κατάστασης των ανθρώπων αυτών. Και αυτό δεν εγγράφεται στη λογική της, την παρούσα των κρατικών ενισχύσεων. Πρέπει δηλαδή να μην να καθίσουμε δυνατόν, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τώρα με επενδύσεις στις περιοχές αυτές για να προλάβουμε την επιδείνωση. Και γι' αυτό πρέπει να ξανασκεφτούμε τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Η διαδικασία αυτή ξεκινάει τώρα οι υπάρχοντες κανόνες ισχύουν μέχρι το τέλος του ερχόμενου έτους. Μπαίνουμε λοιπόν σιγά σιγά στη φάση όπου συζητούμε ε, στην τροποποίηση, για την τροποποίηση των κανόνων αυτών και εδώ εμείς πρέπει να παίξουμε το δικό μας ρόλο και ελπίζω η Επιτροπή να δεχθεί το γεγονός ότι θα πρέπει να αλλάξουν αυτοί οι κανόνες τώρα. Τα μηνύματα που έλαβα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ενθαρρυντικά. Είχαμε μια πολύ καλή ανταλλαγή απόψεων με ε, την Επίτροπο Κεσού που είναι τώρα μέλος της Επιτροπής σας. Ε, υπάρχουν και άλλες φωνές βέβαια στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Ε, έχουμε λοιπόν δουλειά μπροστά μας για το θέμα αυτό και θα, πραγματικά θα ήμουν ευγνώμων αν μας υποστηρίξετε και από αυτού. Δεν θέλω τώρα να μπω σε άλλες λεπτομέρειες, να πω ακόμα κάτι. Ένα από τα ζητήματα που προκύπτουν είναι το πεδίο εφαρμογής, το πεδίο που θα καλύπτει αυτό το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Θα αφορά τις περιοχές ε, ε παραγωγής άνθρακα, 41 περιοχές ε, στην Ευρώπη, έτσι, ε, στην Ανατολική Ευρώπη, στο Νότο, ε, στην Κεντρική Ευρώπη, δεν είναι συζήτηση δηλαδή εδώ παραθεση δηλαδή, Ανατολής Δύσης, αφορά το σύνολο τη Ευρώπη. Ποιο θα είναι όμω το πεδίο, αυτό είναι το ζήτημα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είναι αρκετά περιορισμένο το πεδίο. Πρόκειται για μια πολιτική απόφαση η οποία αφορά τον άνθρακα. Μιλάμε για θέσεις απασχόλησης και παραγωγή που συνδέεται άμεσα με τον άνθρακο, άνθρακα και αυτό πρέπει να είναι η βάση για το ταμείο. Ξέρω ότι υπάρχουν και άλλες απόψεις βεβαίως, αλλά πιστεύω ότι μια στενή εφαρμογή, ένα στενό πεδίο ε, είναι και μια πιο λογική προσέγγιση, διότι για άλλες ε, μεταλλάξεις, μετατροπές που λαμβάνουν χώρα έχουμε ήδη μέσα και δεν πρέπει εδώ να τα μπερδέψουμε. Ήθελα να το πω αυτό εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας και να συζητήσω την ομοδότησή μου μαζί σας ε, και σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που μου δώσατε την ευκαιρία να την παρουσιάσω εδώ στην Επιτροπή σας. Ευχαριστώ πολύ. Euh, Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση αυτή. Ήταν πάρα πολύ σαφής. Μας παρουσίασε ξεκάθαρα πόσο κατεπήγον είναι το πολιτικό ζήτημα στην πραγματικότητα. Πρέπει οπωσδήποτε να δοθούν άμεσα απαντήσεις ε, στα ζητήματα που θίξατε. Θα ήθελα να πω στους συναδέλφους ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έπρεπε να παρουσιάσει την πρότασή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Δεκέμβριο, την ανέβαλε για τον Ιανουάριο. Και αυτή τη στιγμή γίνονται διάφορε διαβουλεύσει και διαπραγματεύσει σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακριβώ για τα ζητήματα κλειδί που μόλι ε, θίξατε εσεί στην παρουσίασή σα. Εμεί εδώ στην συνεδρίαση τη Επιτροπή Ρέτζι ε, συζητάμε και μας ακούνε. Οπότε μας ενδιαφέρει να ακούσουμε τις απόψεις των διαφόρων πολιτικών ομάδων και των διαφόρων μελών της Επιτροπής μας ώστε να διαβιβάσουμε στην Κομισιόν αυτές τις απόψεις διότι ε, επί ενός είμαστε όλοι σύμφωνοι επί του στόχου όπως είχα πει στη διασκέψη υψηλού επίπεδου στην Επιτροπή των Περιφερειών και σε ευχαριστώ και πάλι που με καλέσατε Πρόκειται για μια επανάσταση. Επίκειται δηλαδή μια επανάσταση. Ο στόχος αυτός ε, ε, της εγκατάλειψης των ε, πηγών ενέργειας ε, μας βρίσκει όλους σύμφωνους. Το θέμα είναι αυτό το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Πρώτα απ' όλα πιστεύω πρέπει να ξεχάσουμε την ιδέα που σχημάτισαν πάρα πολύ κάποια συγκεκριμένη στιγμή ότι το ταμείο αυτό συμπεριλαμβάνει τα πάντα, την έρευνα και ένα σωρό άλλα πράγματα και θα χρειαζόμασταν 200-300 δις. Τέτοια θέματα θα ρυθμιστούν αλλού, ίσως στο νέο Green Deal. Αυτό το Ταμείο για τη Δίκαιη Μετάβαση και η σχετική νομοθεσία ζητήθηκαν αρχικά για να μετριαστούν οι οικονομικές, κοινωνικές ε, επιπτώσεις και οι επιπτώσεις στην απασχόληση σε περιοχές οι οποίες ε, υλοποιούν αυτή την ε, ε, μεταβολή. Τις περιοχές δηλαδή που παρήγαγαν άνθρακα. Το κοινωνικό και κοινωνικό το κοινωνικό και οικονομικό κόστος θα είναι τεράστιο πράγματι. Αυτή τη στιγμή η Κομισιόν καλύτερα να λάβει διάφορες αποφάσεις. Εμείς ε, θέτουμε διάφορα ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα είναι αυτό του ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Πρέπει να αφορά μόνο τις περιοχές παραγωγής ε, άνθρακα, τις 41 αυτές περιοχές ή μήπω είναι προτιμότερο να είναι ευρύτερο, να καλύπτει δηλαδή το σύνολο των κρατών μελών με κριτήρια που θα διοχετεύουν τα κονδύλια αυτά προς ε, τις αντίστοιχες περιοχές ε, και κριτήρια που θα επιτρέπουν τη δίκαιη ε, κατανομή. Αυτό είναι ένα πρώτο ερώτημα. Και βάσει αυτού του ερωτήματος θα γίνει εν ευθέτω χρόνο η συζήτηση εδώ στην Επιτροπή μας. Αλλά πιστεύω ότι πολύ συμφωνούμε. αλλά υπάρχουν και αρκετές διαφωνίες για το ζήτημα αυτό. Υπάρχουν περιοχές, υπάρχουν περιοχές που δεν είναι ε, περιοχές παραγωγής άνθρακα, αλλά που εξαρτώνται από τις ενέργειες που παράγονται από ρηκτές πηγές και λένε ότι και αυτές θα υποστούν κάποιο κόστος λόγω αυτής της ε, μετάβασης, αυτής της αλλαγής. Το δεύτερο ερώτημα, ε, και δώσετε εσείς την απάντηση για την Επιτροπή των Περιφερειών, είναι το κατά πόσο οι λειτουργικοί κανόνες της συνοχής πρέπει να εφαρμοστούν στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Η δική μου προσωπική άποψη, αλλά φυσικά δεν είναι άποψη της Επιτροπής μας, η προσωπική μου άποψη είναι ίδια με τη δική σας. Πράγματι πιστεύω ότι οι κανόνες της συνοχής ε, πρέπει να εφαρμοστούν εδώ σε αυτή την περίπτωση. Εκεί τίθενται διάφορα ερωτήματα. Υπάρχει το, ζήτημα, το ερώτημα της χρηματοδότησης, αυτό το ταμείο θα χρηματοδοτηθεί μέσω των ταμείων συνοχής ή θα πρόκειται για νέους πόρους ή για ιδίους πόρους ή για πόρους άλλους που θα ληφθούν από άλλα μέρη του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και εκεί ακόμα δεν έχουν δοθεί ακόμα οι απαντήσεις που χρειάζονται θα δώσω το λόγο τώρα στους συναδέλφους που θέλουν να μιλήσουν και μετά θα σας δώσουμε ε, το λόγο. κύριε κυρία Κρέλα από τους σοσιαλιστές. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για δύο λόγους ασχολούμαι με αυτό το Ταμείο Δικής μετάβαση. ως ε, συντονίστρια για την ομάδα μου εδώ στη Ρέγκη και εγώ προέρχομαι από τη Σαξονία επίσης. Είναι περιοχή παραγωγή άνθρακα. Έχουμε δύο μέρη όπου παράγεται ενέργεια με λιγνίτη και έχουμε την εμπειρία και της Γερμανικής Επανένωσης. Από τη μια μέρα στην άλλη ξαφνικά ε, έκλεισαν 80-90% των ορυχείων, για καλούς λόγους βέβαια, αλλά ξέρω τι σημαίνει όταν ξαφνικά 55.000 ε, ε, σύντροφοι χάνουν τη δουλειά τους. Ε, ανθρακορίχοι, ξαφνικά 55.000 ανθρακορίχοι χάνουν τη δουλειά τους. Είπατε πολύ σαφώς υπάρχει διαφορά μεταξύ της ανταγωνιστικότητας ε, και της πολιτικής απόφασης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό στο πλαίσιο των συζητήσεων. Εγώ τίνω να πω ότι θα πρέπει να περιοριστούμε στις περιοχές ε, παραγωγής άνθρακα. Ξεκινήσαμε με 5 δισεκατομμύρια και τώρα μας λένε οι φήμες ότι Μπορεί να πάμε μέχρι 100 δις, αλλά 5 δισεκατομμύρια για μία περιοχή, αν σκεφτείτε ότι έχουμε 7 κρατήδια ε, και το καθένα έχει μια τουλάχιστον περιοχή, δεν βοηθάει και ιδιαίτερα. «51 δις και 41 περιοχές, 5 ε, δις και 41 περιοχές» σημαίνει ότι η χρηματοδότηση δεν είναι αρκετή, ενώ η χρηματοδότηση θα έπρεπε να είναι σημαντικότερη. Ελπίζω η πρόεδρος της ε, Κομισιόν πριν ε, μας δώσει την πρόταση να αποκτήσει μια καλή ιδέα για το πώς πρέπει να γίνουν αυτά και όχι απλά να παραμείνει κολλημένη στο σχέδιο Juncker. Χρειάζεται το διπλάσιο και το επταπλάσιο Ελπίζω επίσης ότι και τα κράτη-μέλη θα βρουν έναν τρόπο να βρουν χρηματοδότηση. Δεν χρειάζεται και μεγάλη δημιουργικότητα. Ε, ήδη οι πόροι, όπως και αν έρθει, θα πρέπει να γίνει μια ε, προσφορά προς τις περιοχές αυτές. Δεν μπορούμε να τους πούμε απλά θα κλείσουμε τα, τις εγκαταστάσεις και τα ορυχεία και μετά να δούμε τι θα γίνει πρέπει εκ των προτέρων να είμαστε έτοιμοι να έχει γίνει κάποια προετοιμασία. Διότι όλοι πιστεύω αντιλαμβάνονται πολύ καλά ότι ένας ανθρακορίχος ε, δεν θα μπορέσει ξαφνικά να τραφεί από τον τουρισμό και θα, να πάει στο σε ένα ξενοδοχείο να δουλέψει ως μάγειρα. Ένας ανθρακορίχος χρειάζεται μια κανονική δουλειά ε, σε μια βιομηχανία για παράδειγμα. Εκεί θα πρέπει να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Υπάρχουν αρκετές δυνατότητες. Αυτές τις δυνατότητες λοιπόν για να τις εκμεταλλευτούμε χρειαζόμαστε κάποιο πλαίσιο και έναν προϋπολογισμό. Και δεύτερον δεν μπορούμε να κάνουμε σαν να ε, χρησιμοποιούμε διάφορους κανόνες αρρωγής όπως κάνουμε πάντα στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επιχειρήσεις ε, που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις περιοχές θα πρέπει να αξιοποιήσουν και την ευκαιρία να αναπτύξουν δικά τους προγράμματα ή έργα, ούτω ώστε τους δικούς τους ήδη υπαλλήλου, ε, τους εργαζομένους ε, που έχουν ήδη, να τους δώσουν μια ευκαιρία να κάνουν κάτι καινούριο, να βρουν μια δουλειά αφού κλείσουν τα ανθρακοριχεία και οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής αυτές. Στη διάσκεψη της πλατφόρμας για τον άνθρακα στο Γκέρλιτς ε, ήμουν και εγώ εκεί και εκεί κάτσαν μαζί οι περιφερειές και σκέφτηκαν και είπαν ότι υπάρχουν πολλές προτάσεις, πολλά έργα, αλλά χρειάζεται αυτό το νομικό πλαίσιο και ελπίζω ότι θα το συμπεριλάβει αυτό η Κομισιόν στις προτάσεις ε, και σε όλες τις προτάσεις που θα κάνει για βοήθεια προς αυτές τις περιοχές. Ε, αν τα επεκτείνουμε αυτά και στι άλλε περιοχέ, θα έρθουν τα πράγματα άνω κάτω. Χρειάζεται να επικεντρωθούμε στις, ε, σε αυτά τα πολύ συγκεκριμένα σημεία. Αλλιώ υπάρχει κίνδυνο ε, να δημιουργηθεί χάο. Ίσως αργότερα για άλλους κατεξαίρεση κλάδου, αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να βοηθήσουμε αυτέ τι περιοχέ που θα εγκαταλείψουν τον άνθρακα. Και με την γνωμοδότηση που αναφέρατε εσείς, πολύ συχνά ε, μας βοηθά η συνεργασία ε, μαζί σας και πιστεύω ότι θα μπορούσε να έχει μεγάλη επιτυχία και να βοηθήσουμε να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους ώστε αυτή η ενεργειακή μεταβολή να μπορέσει να γίνει με τη δική μας βοήθεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος ε, Νοβάκοφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. <clears throat> Κύριε Σπάχη, Ξέρω ότι το μέλλον ανήκει στις καθαρές τεχνολογίες, ε, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. και τις τεχνολογίες που προστατεύουν το περιβάλλον. Δεν αμφιβάλλω καθόλου. Ωστόσο η μετάβαση αυτή δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί με το κόστος δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων στον κλάδο του άνθρακα και δεν μιλώ ως απόγονος ανθρώπου που εργαζόταν στα ορυχεία. Τα προγράμματα που προσπαθούν να διαχειριστούν τη μετάβαση 50 χρόνων που απομακρύνονται από την αγορά αυτή δεν θα καταφέρουν να τους κάνουν web designer, φαντάζομαι. Ο συνήθι ύποπτο για τη χρηματοδότηση κάθε καινούργια ιδέα τη Επιτροπής είναι το Ταμείο Συνοχής. Είχαν ξεκινήσει με 5 δισεκατομμύρια, μετά είχαν πάει σε 7. Εχθέ η κυρία Πρόεδρος ανέφερε 100 δισεκατομμύρια. Τώρα, όλα αυτά οδηγούν στο γεγονός ότι οποιοδήποτε άλλο ταμείο, οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα θα είναι πιο ισχυρό με περισσότερους πόρους από το Ταμείο Συνοχής και την Πολιτική Συνοχής. Αν αποφασίσουμε ότι η περιβαλλοντική προστασία είναι ύψης της προστασία, ε, προτεραιότητας, με βρούμε νέους πόρους. σε κάποια κράτη-μέλη και στις πιο καθυστερημένες περιφέρειες θα χάσουμε χρηματοδότηση για καθαρότερο νερό ή για εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού. Δεν μπορεί να είναι αυτό το τίμημα. Και εν πάση περιπτώσει αν το εύρος του ταμείου αυτού είναι τόσο μεγάλο τότε τροποποιεί Ουσιαστικότητα και την πρόταση για το ΠΔΠ και για το CPR. Επιπλέον, δεν είναι τα 100 δισεκατομμύρια που θα έχουμε στην αρχή. Αυτός είναι ο στόχος, ο σορευτικός στόχος της Επιτροπής. Δηλαδή μιλούμε για ένα χρηματοπιστωτικό μέσο. Κάτι σαν το InvestEU. εσείς εκπροσωπώντας τις περιφέρειες, όταν συνομιλείτε με τις περιφέρειες του Άνθρακα, για ανθρώπους που προσπαθούν να ζήσουν τις οικογένειές τους με αξιοπρέπεια, αν πάτε και το σπίτι ότι μην ανησυχείτε, θα κλείσουμε τα ορυχεία, αλλά θα βρούμε χρηματοπιστωτικό μέσο, θα βρούμε, είμαι σίγουρος ότι θα ακούσετε. Άρα, εδώ πρέπει να λαμβάνουμε αποφάσεις που να είναι υλοποιήσιμε, όχι απλώς να γεμίζουν στήλε σε εφημερίδες. Αυτό είχα να σας πω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Αντρέ. Για τους ε, πράσινους, ε, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Σπάιχ που μας παρουσίασε την ε, γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών. Συμφωνώ ότι χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα γιατί ο Αντρέα έχει απολύτω ε, δίκαιο. Δεν μπορούμε αυτά να τα πάρουμε από το CPR. Και είπατε κι εσείς ότι θα παίρναμε πόρους από πιο φτωχές περιφερειές για να τις δώσουμε σε περιφερειές που θα είναι πιο φτωχές. Έχουμε το European Trading Scheme για, την, για τα πιστοποιητικά του διοξιδίου και τα έσοδα αυτών των πιστοποιητικών πάνε στα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη τα χρησιμοποιούν τα χρήματα αυτά όπως νομίζουν, όχι για να αντισταθμίσουν την κλιματική αλλαγή. Γιατί αυτός ήταν ο αρχικός στόχος. Όταν μολύνει κανείς το περιβάλλον, εμείς φορολογούμε αυτή τη δραστηριότητα για να αντισταθμίσουμε τα αποτελέσματα. Αλλά δεν συμβαίνει έτσι. Και αν δούμε το Ταμείο της Δίκαιης Μετάβασης, χρειαζόμαστε και χρήματα για έρευνα, χρειαζόμαστε χρήματα και για άλλες δραστηριότητες αντιστάθμισης. Και αν δούμε ένα μέρος αυτών των κονδυλίων και τροφοδοτήσουμε το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, τότε θα έχουμε επαρκείς πόρους και τότε θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Γιατί αν μείνουμε στα 5 δισεκατομμύρια που έχουμε, αν δούμε και τα, τις ε, συγχρηματοδότησης της Τράπεζας Επενδύσεων κτλ, δεν θα πολλαπλασιάσουν τα κονδύλια, θα μείνουν στα 5. Αν μπορούμε να τα διπλασιάσουμε ή να τα τριπλασιάσουμε με κάποια τρίκ, μπορεί να ακούγεται ωραίο αυτό, αλλά ε, το να μείνουν πέντε δις τα χρήματα είναι αστείο για τα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι περιφέρειες. Ε, ε, συμφωνώ απολύτως με αυτά που λέτε. Πρέπει να έχουμε μια συνεργασία οριζόντια εδώ και να βρούμε περισσότερα χρήματα από το πει. Γιατί βεβαίως τα κράτη-μέλη καθόλου δεν είναι διτεθμένα να πούνε ναι θα δώσουμε περισσότερα χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανταλλαγή λοιπόν των ρήπων, το ETS ή οτιδήποτε άλλο είναι ένας καλός τρόπος. Σας ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος κυρία Ντονάτο για το ID. Ευχαριστώ Πρόεδρε θα μιλήσω Ιταλικά. Ευχαριστώ τον κύριο Σπάιχ για την εισήγησή του. Είναι πολύ σημαντική υποστήριξη στην ε, μετάβαση από την παραγωγή άνθρακα το Ταμείο Δικής Μετάβασης με επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους και νομίζω ότι θα πρέπει να αφορά την μετάβαση όχι μόνο από τον άνθρακα αλλά και από τον χάλιβα, διότι η πραγματικότητα η παραγωγική του άνθρακα και του χάλιβα είναι θεμελιωδέστατες για τις οικονομίες αρκετών κρατών μελών ακόμα σήμερα. Η μετάβαση λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Σε ό,τι αφορά στη χώρα μου, έχουμε πολύ θετικές εμπειρίες όπως στην Σαρδινία όπου είχαμε την μετατροπή των παλαιών ορυχείων άνθρακα με διεθνές έργο όπου έχουν μετατραπεί σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας ε, του αργού ε, πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο και που κοιτάει προς το μέλλον και που αξιοποίησε αυτή τη μετάβαση, αλλά έχουμε και διαφορετικές περιπτώσεις, πιο αρνητικέ. Έχουμε την Ήλβα στο Τάραντο που συζητείται πολύ στα μέσα τελευταίως, όπου έχουμε μια παραγωγική πραγματικότητα του χάλιβα υψηλά ρηπογόνα, ε, αλλά και με οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι το, η σημασία του θέματος που αναλύσατε, που εξετάσατε, με μια αναθεώρηση, επανεξέταση των ε, κρατικών ενισχύσεων είναι υψής της σημασίας γιατί πρέπει να υποστηρίξουμε και την παραγωγική διαδικασία και τις θέσεις απασχόλησης που συνδέεται με αυτήν ώστε να έχουμε πράγματι μια δίκαιη, ισότιμη μετάβαση προς την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και αυτά μπορούμε να τα καταφέρουμε και μέσω εξαιρέσεων ή εν πάση περιπτώσει και άλλων προβλέψεων πέραν της ε, απλής απαγόρευσης των κρατικών ενισχύσεων όπως ισχύει σήμερα. Εμείς θα υποστηρίξουμε λοιπόν κάθε είδους τέτοια νομοθετική προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση που θεωρώ πολύ σημαντική και πολύ επίγουσα θα σας έλεγα. Ευχαριστούμε η Ματίνα Μίχελς για την ε, Γκουε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να πω το εξής. Πρώτα απ' όλα ε, ε, υποστηρίζουμε όλες τις τοποθετήσεις που ακούστηκαν εδώ σήμερα που λένε ότι χρειαζόμαστε νέους πόρους, φρέσκους πόρους. Δεν μπορούμε απλώς να μετακινήσουμε τους υφιστάμενους. Δεύτερον, Πρέπει, είναι αλήθεια, να δούμε το θέμα της μετάβασης και πώς ρυθμίζεται αυτό. Ποιες περιφέρειες πρέπει να επωφεληθούν. Μπορεί κανείς να φανταστεί ότι θα υπάρξει μία περίοδος μετάβασης που θα περιοριζόταν στις 41 αυτές ανθρακοπαραγωγές περιφέρειες και που αργότερα, αν ήταν απαραίτητο, θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλες περιφέρειες. Το άλλο που είναι σημαντικό για μας είναι πώς ορίζει κανείς τη δίκαιη μετάβαση. Δεν μπορεί να είναι απλώς ένα μέσο μονόδρομης κατεύθυνσης προς την επίτευξη κλιματικών στόχων. Πρέπει η δίκαιη μετάβαση να ορίζεται με πλήρη τρόπο ώστε να καλύπτει και ανησυχίες κοινωνικές. Δηλαδή να καλύπτει και άλλες διαστάσεις είναι λοιπόν πολύ σημαντικό πώς ορίζουμε τι σημαίνει δίκαιη μετάβαση. Δεν μπορεί να είναι απλώς οικονομικής χρειάς ή απλώς περιβαλλοντικής χρειάς. Εμείς θεωρούμε ότι πάνω απ' όλα είναι κοινωνική η διάστασή της. Ευχαριστούμε. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα μιλήσω ισπανικά. Ευχαριστώ πολύ και καλωσορίζω τον ομιλητή και τον ευχαριστώ για την εισηγησή του. Ήδη ακούσαμε και από τον Πρόεδρο και από τα μέλη μια εστίαση σχετικά με το ποια πρέπει να είναι αυτά τα κονδύλια, ποιοι πρέπει να είναι οι δικαιούχοι, από πού πρέπει να βρεθούν αυτά τα χρήματα. Από την εμπειρία που έχετε και στη Γερμανία, νομίζω ότι πρέπει να εστιαστούμε σε κάτι που είναι ευθύνη γνωρίζοντας επί πολλά χρόνια ότι ο τομέας αυτός ε, είχε πάψει να είναι ανταγωνιστικός, διατηρήθηκε μέσω συγκεκριμένων πολιτικών και άλλων συμφερόντων, υποστηρίχθηκε, ενισχύθηκε με τη σύμπραξη των πολιτικών κομμάτων δυστυχών, ένας τομέας ο οποίος είχε πάψει να είναι ανταγωνιστικός. Ενώ γνωρίζαμε, μπορούσαμε να προβλέψουμε ότι ήταν ένας κλάδος που δεν μπορούσε πλέον να παραγάγει για το μέλλον νέες θέσεις απασχόλησης. Όμως τον είχαμε βάλει σε τεχνητή αναπνοή όλα αυτά τα χρόνια και αυτό έγινε στην Ισπανία σε πάρα πολλές περιφέρειες, στην Αστούρια, στην ε, Ανδαλουσία. Υπάρχουν πολλοί τομεί στην Ευρώπη που αυτή τη στιγμή ε, σταδιακά πάβουν να είναι ανταγωνιστικοί. Υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται στους τομείς αυτούς και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να ε, πάρει τα διδάγματα της, από το τι συνέβη με τα ορυχεία. Και για άλλους τομείς οικονομίας που θα βρεθούν σε λίγα χρόνια στην ίδια κατάσταση. Γιατί τότε θα συζητούμε πάλι πόσα εκατομμύρια ευρώ των πολιτών, των φορολογουμένων πρέπει να δαπανίσουμε για να διατηρήσουμε στην απασχόλησή της ε, πολύ κόσμο που σωστά ανασυχούν για τις οικογένειές τους και το ε, την απασχόλησή τους, αλλά ε, η περίπτωση των ορυχείων είναι μια περίπτωση αποτυχίας συλλογικότατης και πολιτικής. Βεβαίως και πρέπει να δοθεί λύση για τους εργαζόμενους αυτούς, αλλά πρέπει να λαμβάνουμε και τα διδάγματά μας. Ε, επαναλαμβάνω, σε πολλές περιφέρειες της Ευρώπης χάνουμε ανταγωνιστικότητα και διατηρούμε τεχνητά κάποιους κλάδους παραγωγής της οικονομίας. λόγω ε, πολιτικών ή κομματικών ε, συμφερόντων. Σας ευχαριστώ. Πέντρο Μαρκές. Ο Πέντρο Μαρκές έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω και εγώ κάποιες σκέψεις. Η απαλλαγή από μαρκες άνθρακα έχει ε, βίες, ε, βίο αντίκτυπο οικονομικό και κοινωνικό. Και σίγουρα οι περιοχές ε, παραγωγής άνθρακα είναι αυτές που πλήττονται περισσότερο. Αλλά γενικότερα οι επιπτώσεις θα είναι πολύ ευρύτερες και όχι, δεν θα αφορά μόνο τις περιοχές αυτές. Πρέπει να καλωσορίσουμε το γεγονός ότι από ό,τι φαίνεται είμαστε αρκετά πιο φιλόδοξοι σε ό,τι αφορά το Ταμείο για τη Δίκαιη Μετάβαση σε σχέση με τα που πριν από μερικές μέρες μόλις. Δεν ξέρω λεπτομέρειε πληροφορίε, αλλά φαντάζομαι ότι θα υπάρξει κάποια μόχλευση με κάποια οικονομικά μέσα. Ε, δεν νομίζω δηλαδή ότι θα πάρθει ω διαμαγεία μια απόφαση ε, για ιδίου πόρους που δεν μπορούσαμε να έχουμε ε, για χρόνια και χρόνια. Δηλαδή σίγουρα θα υπάρχει κάποια μόχλευση μέσω των οικονομικών μέσων. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ σε μια εμπειρία ε, την εμπειρία μου ως Υπουργού Συνοχής έως ε, πρόσφατα και ήμουν αρκετά έτσι, διστακτικός στη χρήση αυτών των οικονομικών μέσων μέσω της πολιτικής συνοχής. Να σας δώσω ένα παράδειγμα όμως. Εμείς μπορέσαμε, ακόμα και στις πιο φτωχές περιοχές της χώρας, να προσελκύσουμε ιδιωτικέ επενδύσεις, να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης μέσω νέων οικονομικών εργαλείων, μέσων. Εγώ στην αρχή ήμουν διστακτικός, αλλά το κάναμε. Θέλησαμε να φανούμε πιο φιλόδοξοι στι περιοχέ αυτέ. Είπαμε ότι έχουμε αυτά τα χρήματα που θέλουμε να μοχλεύσουμε. Θα πρέπει να περάσουμε από τα κατάλληλα οικονομικά εργαλεία και τα καταφέραμε. Όταν λοιπόν για project τα οποία έχουν μέλλον ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μέσα. Να σας πω λοιπόν, με βάση αυτό το παράδειγμα, ότι μπορούμε να είμαστε λιγότερο αμυντική από την πλευρά μας, από την πλευρά της πολιτικής συνοχής και αυτό θα μας βοηθήσει να υπερασπιστούμε την πολιτική συνοχής ε, στη συνέχεια. Αυτή η παραδοσιακή πολιτική δηλαδή μπορεί να εξχρονιστεί μέσω αυτών των μέσων για τέτοιου ε, ε, επενδύσεις. Βεβαίως υπάρχουν κοινωνικές επενδύσεις, εκεί είναι άλλη ιστορία. Υπάρχουν ε, και άλλες μορφές επενδύσεων που δεν, δεν μπορούν να περάσουν από αυτά τα σύγχρονα μέσα μόχλευσης. Τι συζητάμε εδώ όμως. Θέλουμε κάποια χρήματα της πολιτικής συνοχής να τα διαθέσουμε σε κάποιες περιοχές ή για κάποια project. Διότι έτσι όπως αντιλαμβανόμαστε εμείς αυτό που συζητείτε, τα χρήματα αυτά, μέρος από τα χρήματα, το θα προέρχεται από την, από την πολιτική συνοχής και θα το ονομάζουμε δίκαιη μετάβαση, αλλά θα είναι χρήματα τη πολιτική συνοχή. Οι στόχοι άλλωστε για την ε, απαραγή από τον άνθρακα ε, εντάσσονται στην πολιτική συνοχή. Αν μιλάμε λοιπόν για κάποια χρήματα που θα ε, αφιερώσουμε από την πολιτική συνοχή εκεί, γιατί δεν το λέμε αυτό για περιφέρειες ή για χώρες ε, σε ό,τι αφορά την κεντρική διαχείριση. Γιατί είναι αδύνατο να μιλήσουμε και να, να προέλθουν χρήματα από τις κεντρικές πολιτικές. Για αυτούς τους στόχους. Γιατί λένε να το παίρνουμε τα χρήματα της πολιτικής συνοχής. Αυτό δεν, δεν μπορεί να γίνει αποδεικτό. Αν θέλουμε ένα μείγμα όπου τελικά ε, επιτυχάνονται οι στόχοι μας, αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο μέσω της πολιτικής συνοχής, ε, μέσω των θεματικών μας στόχων. Και οι κεντρικές πολιτικές πρέπει να συνεισφέρουν. Αυτές οι περιοχές ε, που έχουν πληγεί περισσότερο ε, από αυτήν την διαδικασία. Θα πρέπει να γίνουν ανταγωνιστικέ σε άλλους ε, τομείς. Έρευνα, ας πούμε. Πρέπει λοιπόν να περάσουμε και στις κεντρικέ πολιτικέ. Βεβαίω για κάποια θεσμικά όργανα αυτό είναι κάτι το οποίο ούτε κάθε να το συζητήσουμε. γιατί πολιτική συνοχή πάντα λέμε εντάξει, ναι, θα βρούμε χρήματα από εκεί. Ε, ήθελα να το πω λοιπόν αυτό. Εγώ δεν συμφωνώ πρέπει να έχουμε ένα μείγμα πολιτικών και μέσων, όχι μόνο ένα, και όχι πάντα να τα παίρνουμε από την πολιτική συνοχή για να πετύχουμε τους στόχους μας. Πιστεύω ότι ακολουθούμε το σωστό δρόμο, εάν θέλουμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι σε ό,τι αφορά αυτό το Ταμείο Δίκης Μετάβασης, αυτό είναι θετικό, διότι δεν μιλάμε εδώ μόνο για 41 περιοχές, μπορεί να είναι το πρώτο βήμα. Σημαντικό βέβαια ε, το βήμα για αυτές τις περιοχές, αλλά ο στόχος είναι ευρύτερο. Και κάτι τελευταίο, Πρόεδρε. Δεν μπορούμε να πετύχουμε το στόχο της απλαγής από τον, άνθρακο, από τον άνθρακα μόνο εντός των εδαφών μας. Έτσι. Είναι το θέμα των συνόρων. Εισάγουμε άνθρακα μαζικά. Εάν δηλαδή εμείς περιοριστούμε στα σύνορά μας και δεν μιλήσουμε για άλλα πράγματα, όπως φορολόγηση του άνθρακα στα σύνορα, ε, τότε ούτε θα απαλλαγούν από τον και ε, θα πληγούν οι επιχειρήσει μα. Ένα τομέα που χρειάζεται στη χώρα μου, ο τομέα τη αεροπορία. Ναι, παράγουν πολλέ εκπομπέ στα αεροπλάνα, είναι αλήθεια. Εκπέμπουν. Αλλά αν κάνουμε κάτι ε, στα δικά μα όρια, φορολογώντα και δεν κάνουμε τίποτα εκτό συνόρων, στην πραγματικότητα γίνονται πιο ανταγωνιστικέ ε, οι εταιρείε από τη Μέση Ανατολή, παραδείγματο χάρη. Και χάνουμε βεβαίω θέσει απασχόληση εντό συνόρων. Ε, θα πληγεί ο τουρισμό, η αεροπορία. Ε, και αυτοί αγοράζουν καύσιμα στην τιμή του νερού εκεί, έτσι. Λοιπόν, ναι, απαλλαγή από την άνθρακα εντό και εκτό. Ιδάλω οι περιοχέ μα θα υποφέρουν ακόμα περισσότερο. Μάλιστα, ευχαριστώ. Νομίζω ότι ανέφερες όλα τα ζητήματα. Ε, εγώ συμφωνώ μαζί σου. Μόνο με ένα μείγμα μπορούμε να προχωρήσουμε. Βεβαίως ε, αναμένουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όμως με βάση τις δηλώσεις που έγιναν χθες, από ό,τι φαίνεται ο θα είναι σημαντικός, Οπότε προφανώς θα υπάρξει και κάποιο ποσοστό χρηματοδότησης, ε, προφανώς και θα υπάρξουν κάποια οικονομικά μέσα, δεν ξέρω, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, InvestEU ε, και χρήματα βεβαίω στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Σίγουρα θα αποτελέσει σε ένα προϊόν ενό μείγματο, εν αυτή η προσπάθεια. Εφόσον μιλάμε για κάτι βεβαίω πολύ πιο μεγάλο και όχι απλά 5 δις Λοιπόν, Ροντρίγκε Ράμος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η συζήτηση αυτή είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και είναι και επίκαιρη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή είναι στην COP25 στη Μαδρίτη και ηγείται μιας προσπάθειας, μιας διαδικασίας μετάβασης προς ένα σύστημα ε, καθαρής ενέργειας που δεν θα μολύνει. Η φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2050 να είμαστε ε, ουδέτεροι σε επίπεδο εκπομπών ενεργειακών ε, νομίζω πως είναι ένα δείγμα το ότι είμαστε στην πρώτη γραμμή και βεβαίω η ευημερία των συμπολιτών μας, η μελλοντική, παίζεται τώρα, σήμερα. Ε, κατά πόσο θα μπορέσουμε με έξυπνο τρόπο αλλά και με θάρρος να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία ε, μετάλλαξης, ε, μετασχηματισμού ε, σε ενεργειακό επίπεδο. Βεβαίως ε, όλοι, όλες οι περιοχές θα πληγούν, αλλά οι περιοχές εκείνες όπου η οικονομία, του, η οικονομία εξαρτάται ή εξαρτιόταν στο παρελθόν από την εξορίξεις άνθρακα, εκεί προφανώς βραχυπρόθεσμα οι επιπτώσεις θα είναι σκληρές. Δεν είναι μόνο η παραγωγή, η εντατική του άνθρακα, είναι και όλη η οικονομική δομή, η επικουρική ε, που εξαρτάται από αυτή τη δραστηριότητα ή εξαρτιόταν από αυτή τη δραστηριότητα. Πέρα λοιπόν από τα ερωτηματικά που τέθηκαν στη σημερινή συζήτηση, αλλά και στο έγγραφο της Επιτροπής των Περιφερειών, χώρες όπως η δική μου, η Ισπανία, με σημαντικές περιφέρειες που επηρεάζονται και η δική μου αυτόνομη περιφέρεια, η Καστήλη και Λεόν, όπου είχαμε τέτοιες ε, εξορίξεις οι οποίες σταμάτησαν. Γνωρίζουμε ότι είναι πολύ δύσκολο. Αυτό λοιπόν είναι το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης που θέλει βραχυπρόθεσμα να μην βρεθεί κανένα ευρωπαίος πολίτης μόνος του ή να μην μείνει πίσω, θα πρέπει να περιλαμβάνει το ταμείο αυτό και τις περιοχές εκείνες που ήδη έχουν ξεκινήσει μια διαδικασία ενεργειακής μετάβασης που έχουν δηλαδή ήδη ολοκληρώσει ε, το κλείσιμο κάποιων ορυχείων και που πολύ μεγάλες δυσκολίες σε αυτή τη διαδικασία ε, οικονομικής και κοινωνικής ε, δομικής μετάβασης στις περιοχές τους. Ξέρετε ότι είναι μακροπρόθεσμα, είναι μια διαδικασία η οποία κοστίζει πολύ. Το γεγονό ότι έχουν ή δεν έχουν πλέον ορυχεία, αν τα έχουν κλείσει πρόσφατα ή όχι, δεν θα πρέπει να είναι κριτήριο. Η αναγκαιότητα πάντως οι πολίτες ε, να δουν ότι υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές συνοδευτικές ε, σημαίνει ότι αυτή η κοινωνική μετάβαση είναι απαραίτητη. Το νέο σύστημα παραγωγής και σε ό,τι αφορά τι μεταφορέ, ό,τι αφορά την ενέργεια, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια μεγάλη επένδυση σε τομέα καινοτομία, των νέων γνώσεων. Αλλά βεβαίως, βραχυπρόθεσμα θα πρέπει να βοηθήσουμε του εργαζόμενου και τι εργαζόμενε αυτού και να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στους κλάδους εκείνους που θα πληγούν περισσότερο από τις επιπτώσεις αυτής της διαδικασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Ζολιβό. Uh, thank you very much. συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ έχω εργαστεί σε μια από τις φτωχότερες περιοχές ε, της Βορειάς Αγγλίας, μια μικρή-μικρή κομιτεία με μια πολύ φτωχή κοινότητα. Ο άνθρακας ήταν οικονομική βάση για όλη την κοινοτική και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο για όλα αυτά που συζητάτε σήμερα, διότι εκεί δεν υπήρχε τίποτα ε, στις κοινότητε με τις οποίες εγώ εργαζόμουν, όχι μόνο άνθρακα, υπήρχε και χαλιβουργία εκεί στο Κάντιντορν. Το να αντικαταστήσει αυτές τις βιομηχανίες ε, με μια βιομηχανία chips, ε, γιατί αυτό συνέβη, δεν λύνει τα προβλήματα. Μιλάμε για δουλειές για τους ανθρώπους, για τις οικογένειές τους, για την αξιοπρέπειά τους η οποία καταστράφηκε από το γεγονός ότι δεν τους δόθηκαν ποιοτικέ θέσει εργασίας όπου να μπορούν να αξιοποιήσουν τις ε, εξαιρετικές τους ικανότητες σε θέματα μηχανικής. Τον εργάζονται τελικά σε κάποια βιομηχανία παραγωγής ε, πακέτων chips ε, και εκεί να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες τους αντί για την εξόρυξη ανθράκα. Όλα αυτά κατέστρεψαν ακόμη και την αισθήση αλληλεγγύη που αισθάνονταν μεταξύ τους, ε, κατέστρεψαν την αξιοπρέπεια που αισθάνονταν και ακόμα δεν έχουν ε, ε, περάσει αυτά τα τραύματα. Δεν χρειάζονται απλά νέες δουλειέ, χρειάζονται δουλειέ νέες, καλή ποιότητα που να αναγνωρίζουν τη συμβολή αυτών των εργαζομένων, αυτών των ανθρώπων στην κοινωνία μας ε, για να τους δοθεί η αξιοπρέπεια που χρειάζονται για να βοηθηθούν να συνεχίζουν να κερδίζουν το ψωμί που χρειάζονται οι οικογένειέ του. Γιατί αλλιώ καταλήγει κανεί σε μια κατάσταση όπω αυτή που έχουμε τώρα. Πρέπει να σα πω σε, κατά σε ενίες, ε, κατά μία έννοια, το Brexit είναι η απάντηση σε αυτό. Οι ξεχασμένε κοινότητε ε, του άνθρακα στη Βόρεια Αγγλία, όταν η Μάργαρετ Θέτσερ του εγκατέλειψε κλείνοντα τα ορυχεία χωρί να τα αντικαταστήσει με τίποτα. Αυτό το τίμημα πληρώνουμε τώρα. Έχουμε κάποιες άριστες πρωτοβουλίες, ε, το καταπίστευμα για την αναγέννηση των ε, περιοχών άνθρακα, το οποίο κάνει καταπληκτική δουλειά. Πιστεύω ότι η σημερινή συζήτηση είναι πολύ σημαντική για το μέλλον της Ευρώπης και για τις εκατοντάδες χιλιάδες ε, εργαζομένων ανθρώπων, απλών ανθρώπων που ξέρουν ότι δεν θα τους ξεχάσουμε. Εγώ υποστηρίζω το νέο πράσινο σύμφωνο, δεν θέλω τον άνθρακα, αλλά δεν μπορούμε να ξεχνάμε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Η δίκαιη μετάβαση πρέπει να σημαίνει κάτι στην πραγματικότητα. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμβολή σας. Είναι μια διάσταση πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ σημαντική για τη συζήτησή μας στο μέσα Μαρτίν Ντεαλμάγο, έχετε το λόγο. Eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ευχαριστούμε και τον κύριο Σπάιχ. Ήθελα να ξανααναφέρω κάτι που ήδη σχολιάστηκε, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Για την δυνατότητα ή και τον κίνδυνο υπό τη δική μας οπτική, κάποιες ε, κομιτείες, κάποιες ε, περιφέρειες να μείνουν εκτός της κάλυψης αυτού του Ταμείου της Δικαίης Μετάβασης. Και εκείνες οι χώρες και εκείνες οι περιφέρειες που έκαναν τη δουλειά τους, έκλεισαν τα ορυχεία, εκτέλεσαν το καθήκον τους αλλά ξαναβρίσκονται σε ένα περίπλοκο πλαίσιο κοινωνικής και εργασιακής μετάβασης μπορεί να μείνουν εκτός της κάλυψης των πόρων αυτών, των κονδυλίων αυτών. Ενώ εκτέλεσαν τα καθήκοντά τους πλήρως και πολύ πρόσφατα ολοκλήρωσαν. Επομένως, τι εννοούμε περίοδο μετάβασης χρονικά. Ποια είναι μια δίκαιη χρονική περίοδος μετάβασης ώστε να προσφερθεί μια, εναλλακτική, μια ποιοτική εναλλακτική για την απασχόληση των ανθρώπων αυτών. Έχω την ε, εντύπωση, μάλλον έχω την ανησυχία ότι οι περιοχές αυτές που κατάφεραν να κάνουν αυτήν την ε, να ολοκληρώσουν τη διαδικασία κλεισίματος των ορυχείων δεν θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτά τα υπόλοιπα της μετάβασης έτσι όπως τίθενται τα όρια της περίοδου αυτής. Χρειάζεται η προστασία του περιβάλλοντος, αλλά μπορεί, επαναλαμβάνω, κινδυνεύουμε να μείνουν οι περιοχές αυτές εκτός της, της, της περίοδου έτσι όπως την ορίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Τελευταία ομιλήτρια η Μαρία Σπυράκη. Thank you, Chair. Thank you, Mr. Spike, for having you here. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε κύριε Σπάκη που ήρθατε εδώ στο Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να υπενθυμίσω αρχικά την περσινή μα συνάντηση, το, συγγνώμη, το περασμένο καλοκαίρι, όταν συζητήσαμε ότι το Ταμείο Δίκαιης μετάβαση ε, θα χρηματοδοτηθεί με διάφορου τρόπου. Ε, αυτό συζητήσαμε και επιμένω ε, θα πρέπει να έρθουν κονδύλια από το νέο πολιτή δημοσιονομικό πλαίσιο ώστε να υπάρχει μια σταθερή χρηματοδότηση. Φυσικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επιπλέον χρηματοδότηση για τι περιοχέ που εξαρτώνται από τον άνθρακα είτε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, είτε από τον ιδιωτικό τομέα, είτε από του εθνικού προπολογισμού. Αλλά είναι σημαντικό να υπάρχει μια σταθερή βάση ω αφετηρία. Δεύτερον, θα ήθελα να κάνω κάποιε ερωτήσει όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί το Ταμείο Δίκαιης μετάβαση όταν θα ξεκινήσει τη λειτουργία του. Πρώτον, η βάση τη ε, απαλλαγή από τον άνθρακα στην χώρα μου, στην Ελλάδα, η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει όλα τα εργοστάσια άνθρακα μέχρι το 2028. Είναι πάρα πολύ γρήγορη η απαλλαγή αυτή των άνθρακα. Πολύ γρήγορη μετάβαση. Ειδικότερα όσον αφορά περιοχές όπως η Δυτική Μακεδονία που εξαρτάται από τον άνθρακα ε, πλήρως. Το 45% του τοπικού ΑΕΠ προέρχεται από τον άνθρακα, από το λιγνίτη και για την περιοχή της Μεγαλόπολης που είναι ανήκει στην Πελοπόννησο. Η απαλλαγή από τον άνθρακα είναι ένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας ε, για χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Η διαδικασία επιλεξιμότητας είναι πολύ σημαντική για αυτή την περιοχή, ειδικότερα για τη Μεγαλόπολη, η οποία δεν είναι περιφέρεια ολόκληρη, είναι ένα μικρό κομμάτι της Πελοποννήσου. Δεύτερον, ήθελα να πω δύο λόγια για τους ανθρώπους που εργάζονται στο λιγνίτη, με, το λιγνίτη, με τον άνθρακα και τους ανθρώπους που σχετίζονται με όλα αυτά ε, με τους ανθρακορίχους, ε, ε, με τους εργαζομένους στο λιγνίτη, στον άνθρακα. Πρέπει να εστιαστούμε σε αυτούς γιατί είναι μεσήλικες και πρέπει να τους διευκολύνουμε να μετεκπαιδευτούν, να αναβαθμίσουν τις ικανότητές τους και ήθελα να πω και κάτι άλλο που προσπαθώ να επαναλαμβάνω διαρκώς. Δεν είναι εύκολο να μετασχηματίσεις έναν ανθρακορύχο σε εμπειρογνώμονα σε κάποιον άλλο κλάδο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ Μαρία. Είδατε, ήταν πολλές ερωτήσεις, η συζήτηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Τώρα ξεκινά ουσιαστικά. Αλλά η Επιτροπή μας είναι έτοιμη να ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό. Σας δίνω το λόγο για να απαντήσετε στο σύνολο των ερωτήσεων που σας ε, τέθηκαν. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτον, σας είμαι ευγνώμων για τα ενθαρρυντικά σας λόγια. Μου δείχνετε ότι η πρωτοβουλία μας βρίσκεται στο σωστό δρόμο, αλλά φυσικά τέθηκαν κάποια ζητήματα, στα οποία θα ήθελα να απαντήσω. Ένα πράγμα που θέλω να τονίσω, ίσως να μην το ανέφερα, να μην το ανέλησα επαρκώς στην αρχική μου παρουσίαση, υπάρχει μια σαφής διάκριση μεταξύ της εγκατάλειψης του άνθρακα για λόγους ανταγωνιστικότητας και της εγκατάλειψης του άνθρακα για λόγους πολιτικούς για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Θα ήθελα λοιπόν να συνενώσουμε αυτές τις δύο προοπτικές, αυτό που ακούσαμε για την Ισπανία και την προοπτική της Αξονίας στη Γερμανία. Γιατί στη Σαξονία μιλάμε για λιγνίτη. Ο λιγνίτης είναι μια φθηνή μορφή ε, παραγωγής ενέργειας είναι στο έδαφος, ε, κοντά, ε, μπορεί να γίνει εξόρυξη φθηνά και είναι πολύ ανταγωνιστικός. Οπότε οι δουλειέ αυτέ αξόνια αμείβονται πάρα πολύ καλά. Η βιομηχανία είναι πάρα πολύ σύγχρονη, έχει εξυγχρονιστεί πλήρω. Οι άνθρωποι που εργάζονται και οι οικογένειε που ζουν από αυτό έχουν προοπτικές για πολλές δεκαετίες αν δεν είχε ληφθεί η πολιτική απόφαση εγκατάλειψη του λιγνίτη. Στη δική μα περιοχή έχουμε και τα δύο. Και το λιγνίτη που είναι ανταγωνιστικό και τον άνθρακα που είναι ε, ε αντικείμενο επιχορήγηση, τεράστιων επιχορηγήσεων και συμφωνώ. ίσως χρειάστηκε πολύ καιρό η διαδικασία του να περάσουμε από αυτή τη μορφή ενέργεια σε, ε, άλλε πηγέ ε, εσόδων. Έγινε, Έγινε μέρη για κοινωνικούς λόγους, για να παραμείνουν οι άνθρωποι στα ορυχεία γιατί δεν υπήρχε εναλλακτική. Και πληρώσαμε ένα τεράστιο τίμημα γι' αυτό. Αλλά ήθελα να έχετε υπόψη σε αυτή τη διάκριση. Πολλοί από εσάς ε, θεξάτε το ζήτημα του τι θα κάνουν οι άνθρωποι που εργάζονται τώρα στα ανθρακοριχεία ε, ή σε σχετικές ε, θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τον κύριο Νόβακοφ και την κυρία Ward, ένα αφηρημένο πρόγραμμα δεν βοηθά κανέναν. Με τέτοια αφηρημένα προγράμματα, όταν πας να τα εφαρμόσεις έναν 50χρονο, τι προοπτικές να του δώσεις. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πιστεύω η σχέση με την πολιτική συνοχή είναι τόσο σημαντική γιατί ο μηχανισμό αυτό τη συνοχή μεταφράζει ένα αφηρημένο πρόγραμμα σε μια συγκεκριμένη πρόταση. Ταυτόχρονα υπογραμμίζει το γιατί χρειάζεται να αλλάξουμε τους κανόνες της κρατικής βοήθειας είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε νέες βιομηχανίες με θέσεις εργασίας σε αυτές τις περιοχές, να βοηθήσουμε την εγκατάσταση αυτών των βιομηχανιών, ενδεχομένως και με κρατικές ενισχύσεις, για να γίνουν πιο ελκυστικές και όχι να προσφέρουμε δουλειές οι οποίες είναι άσχετες και ε, που πλήττουν και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων που εργάζονται στα ορυχεία, να προσφέρουμε ανάλογες, συγκρίσιμες δουλειές ε, όπου μπορούν να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους. Αλλά πρέπει να είμαστε σαφείς ότι η προσέγγιση αυτή έχει δύο πτυχές αφενός. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι αυτές οι περιοχές στις οποίες αναφερόμαστε θα αναπτύξουν τις δυνατότητες, τις πιθανές αλυσίδες αξίες για το μέλλον. Αλλά εδώ μιλάμε για το μέλλον των παιδιών αυτών που εργάζονται τώρα στα ορυχεία. Και εκεί θα πρέπει να γίνει κατάλληλη έρευνα, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι βιομηχανίε αυτές, οι κλάδοι αυτοί του μέλλοντος. Για να το πω έτσι. Δεν είναι απλή η απάντηση για τους ε, ανθρώπου που εργάζονται τώρα στην ανθρακορυχία. Αυτοί χρειάζονται δουλειέ εδώ και τώρα, τι οποίε πρέπει εμεί να πάμε σε αυτέ τι περιοχέ. Είναι δηλαδή διτή αυτή η προσέγγιση και πρέπει να καλύψουμε και τι δύο πτυχέ. Και για τι δύο αυτέ πτυχέ χρειαζόμαστε το Ταμείο Δίκαιη Μετάβαση. Επίση, ήθελα να τονίσω σε σχέση με τα όσα είπε η κυρία Μίχελ, δεν είναι μόνο οικονομικά τα ζητήματα, είναι και κοινωνικά Γι' αυτό η γνωμοδότησή μου ε, λέει η κοινωνικο-οικονομική αλλαγή και το κοινωνικό σκέλος είναι εξίσου σημαντικό. Φυσικά πρέπει να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και μέλλον ε, οικονομικό για αυτούς τους ανθρώπους, αλλά πρέπει και η κοινωνική πολιτική να υπάρχει για να βοηθήσει όσους χρειαστούν τη βοήθεια και για να τους βοηθήσει να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους, τις ικανότητέ τους. Δεν είναι απλά να φέρουμε τους ανθρακόρυφου σε νέες δουλειές, είναι και να αναβαθμίσουμε και τις ικανότητέ του. Πρέπει να είναι πολύ σαφέ αυτό και α μην είμαστε αφελεί. δεν είναι εύκολο αυτό, είναι κάτι πολύ δύσκολο. Και δεν έχουμε όλα τα εργαλεία που χρειαζόμαστε για κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να τα αναπτύξουμε αυτά τα εργαλεία και στον κλάδο τη ε, ε, ε, πολιτικής ε, Φυσικά, ένα από τα βασικότερα ζητήματα ήταν το από πού θα έρθουν τα χρήματα. Εδώ πολλοί συμφωνούν ότι χρειάζονται παραπάνω χρήματα, αλλά από πού θα έρθουν. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Θα εξαρτηθεί από πολιτικές αποφάσεις, σαφώς. Πολύ το αναφέρατε. Και το άκουσα και νωρίτερα στη συζήτηση. Δεν θα τα φέρει ο Βασίλης την πρωτοχρονιά. Φυσικά εγώ δεν γνωρίζω πολύ καλά, γιατί ασχολούμαι σε περιφερειακό επίπεδο περισσότερο. Ίσως θα είναι ένα συνδυασμό νέων πηγών ε, χρηματοδότηση Το ETS αναφέρθηκε εδώ, ίσως και επιπλέον κονδυλίων από τα κράτη-μέλη, αλλά φυσικά δεν ε, αρνούμε ότι είναι πολύπλοκο το θέμα. Και δεν, είπα και εδώ δεν πρέπει να είμαστε αφελεί. Είναι πολύ δύσκολο το θέμα, αλλά δεδομένη τη τεράστια δυσκολία του θέματος της κλιματικής αλλαγής, ε, είμαι πεπισμένος ότι χρειαζόμαστε αυτά τα επιπλέον χρήματα. Κάπου θα πρέπει να βρεθούν. Κύριε Μαρκές, αυτό που είπατε θα πρέπει να το σκεφτώ λίγο παραπάνω. Το να συνδυάσουμε το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης που σχετίζεται στενά με την πολιτική συνοχής με τη δέσμευση χρηματοδοτικών μέσων σε ταμεία κεντρικής διαχείρισης είναι μια πολλά υποσχόμενη ε, οδός χρήση περαιτέρω διερεύνηση. στο να δεσμεύσουμε χρήματα τα οποία αποτελούν το αντικείμενο κεντρική διαχείριση θα μπορούσε να προσφέρει την κατάλληλη υποστήριξη. Οπότε σα ευχαριστώ για την ιδέα. Και φυσικά το εύρο, το αντικείμενο και το είπα ήδη και στην αρχική μου παρουσίαση το εύρο του Ταμείου είναι πράγματι σημαντικό και παρατηρώ ότι κάποιες ε, περιφέρειες και τις περιοχές έχουν ήδη ξεκινήσει την εγκατάλειψη του άνθρακα. Για αυτούς δηλαδή δεν είναι κάτι μελλοντικό, αλλά είναι το παρόν. Και ο λόγος είναι φυσικά η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής ε, και σε αυτό θα χρειαστούν και εκεί βοήθεια. Αν εγκατέλειψαν τον άνθρακα για λόγους ανταγωνιστικότητας, εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και, και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα είναι διαφορετικά για να βοηθήσουμε αυτή τη διαδικασία. Για να σα δώσω ένα παράδειγμα από τη δική μου περιοχή, θα σα έλεγα ότι η εγκατάλειψη του λιγνίτη, διαδικασία που θα ξεκινήσει πολύ σύντομα, κάνει την περιοχή μας επιλέξιμη για το Ταμείο, αλλά η αποχώρηση από τον άνθρακα είναι κάτι που αποκλείω. Διαφορετικά, όπως είπα, θα μείνουν μισό εκατομμύρια άνθρωποι άνεργοι εκεί πέρα με μια σειρά από τελείως διαφορετικά προβλήματα. Αυτή είναι η λογική και για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Εκεί θα χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τις περιοχές που θα πληγούν από αυτές τις νομοθεσίες, από αυτά τα νέα μέτρα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και όχι για περιοχές που πραγματοποιούν την αλλαγή για λόγους ανταγωνιστικότητας. αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολο να διακρίνουμε λίγο ε, την πολιτική βούληση αφενός καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και της ε, βούληση για ανταγωνιστικότητα από την άλλη. Είναι πολύπλοκο, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι κοινωνικο, οικονομικές αλλαγές σε μια περιοχή ε, σχετίζονται στενά με την πολιτική για την κλιματική αλλαγή και αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Και φυσικά δεν είναι μόνο ο άνθρακας το θέμα, είναι και ο Χάλιβας, το είπε η κυρία Ντονάτο. Και εδώ μπορούμε να ε, σχεδιάσουμε νέες μορφές ε, παροχής ενέργειας. Μόλις άνοιξε το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής ε, καύσιμου υδρογόνου στην περιοχή μας, συγγνώμη, παραγωγής χάλιβα χωρίς άνθρακα. Και αυτή η παραγωγή χάλιβα χωρίς άνθρακα είναι κάτι που θα πρέπει να συνεχίσουμε και να το επεκτείνουμε, γιατί χρειαζόμαστε χάλιβα και απλά πρέπει να απαλλάξουμε την παραγωγή χάλιβα από τις ανθρακούχες εκπομπές. Δεν είμαι βέβαιος αν κάλυψα όλα, αλλά νομίζω τουλάχιστον κάποια από αυτά που ρωτήσατε. Και ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά ότι είμαι ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να έρθω εδώ να σας παρουσιάσω αυτή την πρωτοβουλία, αλλά και που βλέπω πόσο συμφωνούμε ενθαρρυντικά θετικά τα μηνύματα που θα πάρω μαζί μου ότι η Επιτροπή Ρέτζι θα αναλάβει τα πράγματα στα χέρια της ε, κατά κάποιο τρόπο και είμαι βέβαιος ότι θα παρακολουθείτε στενά τις διαδικασίες ε, με το Ταμείο δική Μετάβαση στο μέλλον. Σας είμαι ευγνώμων για τις προσπαθίες σας. Ευχαριστούμε αγαπητέ Μάρκ ε, για την συνεισφορά αυτή που είναι πολύ σημαντική για την Επιτροπή μας. νομίζω ότι είναι ασφαλές να πω ότι πάρα πολλά στοιχεία που βρίσκονται στην γνωμοδότησή σας θα βρίσκονται και στην ε, έκθεση της δικής μας Επιτροπής και στην τοποθέτηση δηλαδή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. με βεβαίως τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαστε απολύτως έτοιμοι εμείς ως Επιτροπή να αναλάβουμε τα καθήκοντά μας ως συνομοθέτης επί του κανονισμού αυτού. Υπάρχει βέβαια και ένα σημείο της γνωμοδότησής σας ε, που είναι πολύ σημαντικό, αυτό της προσθετικότητας. Μιλούμε για 40 δισεκατομμύρια ευρώ που θα στοχευθούν προς την προσπάθεια για το κλίμα. Στην περίοδο 14-20. Επομένως έχουμε νέες δυνατότητες μέσω της προσθετικότητας για χρηματοδότηση. Όλοι παρακολουθούμε προσεκτικά ε, την προσπάθεια αντιστάθμισης των κοινωνικών επιπτώσεων εκεί που το πλήγμα θα είναι μεγαλύτερο για την απασχόληση. Στις περιφέρειες δηλαδή εκείνες. Αυτά είχα να πω συνοψίζοντας τη συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ. Εχθές με πολλούς άλλους συναδέλφους γιορτάσαμε τα 25 χρόνια της Επιτροπής των Περιφερειών. Είμαι βέβαιος ότι έχουμε πολύ ωραία χρόνια μπροστά μας και εμείς και εσείς συνεργασίας σας ευχαριστώ και στο επανειδήν. Bien. Nous allons arriver au terme de Λοιπόν, ολοκληρώνουμε, ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων, θα κάνω κάτι ασυνήθιστο, αλλά σήμερα 5 Δεκεμβρίου είναι τα γενέθλια του υπευθύνου του γραφείου μου, του επικεφαλής του γραφείου μου, είναι πολύτιμος ε, για τη δουλειά μου ως πρόεδρος της Επιτροπής. Χρόνια πολλά του εύχομαι. Voilà. Joyeux anniversaire, Olivier. Χρόνια πολλά, Ολιβιέ. Ευχαριστώ όλους. Θα μείνουμε για την Επιτροπή των Συντονιστών. Θα ζητούσα από όλους εκείνους που δεν τους αφορά το θέμα αυτό να εγκαταλείψουν την αίθουσα. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα 5 λεπτών. Ευχαριστώ.